nehmen unsere Beratungen wieder auf und ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Rechnungshof zum nächsten Tagesordnungspunkt noch auf dem Flughafen festsitzt. Καλησπέρα. παρακαλώ. Ο κύριο Ρούσο ίσω έχει καθυστερήσει. Θα λάβει το λόγο μόλι έρθει. Κάποιο πρόβλημα θα αντιμετώπισε. Χαιρετίζουμε και τον κύριο Ζελμάγερ. Καλώ ήρθατε. Χαιρόμαστε που σα βλέπουμε. συχνά ε, έχουμε συζητήσει για σας, μας είστε γνωστός παρότι δεν έχουμε συναντηθεί. Και θεωρούμε ότι αντί να μιλάμε ο ένας για τον άλλον, καλύτερα να μιλήσουμε μεταξύ μας. Θα σας δώσουμε το λόγο κατευθείαν και μετά ο κύριος Ρούσο θα μας παρουσιάσει το κεφάλαιο 10 όταν θα έρθει κοντά μας. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλείτε σήμερα στο πλαίσιο της, διαδικασίας, της Απαλλαγή διαδικασίας απαλλαγής. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, παρότι δεν έχει έρθει ακόμη το ελεγκτικό συνέδριο. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι συμβατό με τα ε, διεθνή λογιστικά πρότυπα και θα προσπαθήσω να ε, ανταποκριθώ στο ρόλο μου, μιας και πρώτη φορά έρχομαι στην Επιτροπή σας. Δεν σας είχα συναντήσει, χαίρομαι που σας γνωρίζω. Τέσσερα τμήματα για τις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Καταρχήν, θέλω να σας πω δύο λόγια για το ρόλο της Γενική Γραμματείας τη Επιτροπής. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε το αντικείμενο που συζητάμε. Δεύτερον, να σας μιλήσω και για τη διαδικασία απαλλαγής για το 2017. Τρίτον, ορισμένα σημεία που θα είναι σημαντικά για τον εισηγητή, για την προστιθέμενη αξία αυτών που κάνουμε τώρα και στους επόμενους μήνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέταρτον πώς προετοιμαζόμαστε για του χρόνου, για το ε, ενδιαφέρον επόμενο έτος το 2019. Πρώτον, ο ρόλος ε, της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής ο Γενικό Γραμματέα τη Επιτροπή λειτουργεί διαφορετικά από ότι ο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο επικεφαλή τη διοίκηση. Αυτό δεν ισχύει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δεκαετία του 50, έχουμε τρει γενικέ λειτουργίε ο πρώτος γενικός γραμματέας, ο Εμίλ Νοέλ, που ήταν το, είναι το μοντέλο για κάθε υπάλληλο της Επιτροπής, ε, είχε καθιδρύσει αυτό το ρόλο. Είμαστε καταρχήν αυτοί που ασχολούνται με όλες τις γραπτές διαδικασίες, όλες τις διαδικασίες του σώματος της Επιτροπής. Περνάνε όλα από τη Γενική Γραμματεία. Δεύτερον, διασφαλίζουμε τη συνέπεια μεταξύ των, των ε, υπηρεσιών της Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας συντονίζει, διασφαλίζει τη συνέπεια, δεν ορίζει, δεν προσδιορίζει και δεν υπαγορεύει ε, στους άλλους αυτά που θα κάνουν, αλλά συντονίζει τις διαδικασίες της Επιτροπής. Και τρίτον, διασφαλίζουμε ε, τις ομαλές ε, διοργανικές σχέσεις με τα άλλα όργανα, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών και τα Εθνικά Κοινοβούλια δρούμε υπό την αιγίδα του Προέδρου, βοηθούμε τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του και κατά την Προεδρία Γιούγκερ υποστηρίζουμε και τι λειτουργίε του Αντιπροέδρου. Δεν έχουν υποστηρικτική υπηρεσία. Η Γενική Γραμματεία τη Επιτροπή είναι η υποστηρικτική υπηρεσία και για τον ε, Αντιπρόεδρο. Δεν είμαστε λοιπόν υπεύθυνοι για την πληροφορική, δεν είμαστε υπεύθυνοι για άλλα θέματα όπω είναι ο, Γενικό του, ο του Κοινοβουλίου. Εμεί συντονίζουμε τι λειτουργίε, αλλά ε, δεν είμαστε υπεύθυνοι. Είμαστε απλώ υπεύθυνοι για τη συνοχή όλων των πολιτικών. Τώρα δύο λόγια για τη διαδικασία απαλλαγή του 2017. Νομίζω ότι από τον Επίτροπο Έτιγκερ και τους άλλους επιτρόπους θα έχετε ακούσει όλα αυτά. Θα συνοψίσω αυτά τα οποία ήδη γνωρίζετε και ήδη έχετε διαβάσει. Είμαστε στο 11ο έτος που το, Συμβούλιο, το ηλεκτρικό Συνέδριο ε, διαπιστώνει ότι είναι ειλικρινή και οι λογαριασμοί. Ε, το ε, σφάλμα έχει μειωθεί σε ένα ελάχιστο επίπεδο. Είμαστε στο 2,4% που είναι το καλύτερο ποσοστό που είχαμε ποτέ. Βελτίωση λοιπόν και κάτι που μπορεί να επιβεβαιώσει και το ε, ελεγκτικό συνέδριο είναι ότι δεν υπάρχει ουσιώδες φάλμα. Είμαστε ε, ε, υπερήφανοι και είναι και αυτονόητο ότι θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ε, για βελτίωση. Και αυτό να το έχετε κατά νου όταν ε, διαπραγματευόμαστε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό που θέλουμε είναι ο ε, προϋπολογισμός να αντιπροσωπεύει την αξία που έχουν τα χρήματα των φορολογουμένων και θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή είναι σύμμαχος με το Ελεγκτικό Συνέδριο και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση στην εκτέλεση του προϋπολογισμού θα έχετε δει ότι η προστιθέμενη αξία και η απόδοση είναι τα βασικά στοιχεία στι προτάσει μα για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, τι προτάσει που παρουσίασε η Επιτροπή τον ε, Μάιο και τον Ιούνιο και όπου καταβάλουμε συνεχώ προόδου, ακόμη και ε, απρόσμενε προόδου στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τώρα, μια και μίλησα για την απόδοση, να πω δύο λόγια ε, και για την προστιθέμενη αξία. Τι έχουμε κάνει με τον προπολογισμό, με τους πόρου τη Επιτροπής, εστιάζοντας και στα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα. Τονίζω, καταρχήν, τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δημιούργησαν αυτή τη διαδικασία μετά την εμπειρία που είχαμε με την δημοσιονομική κρίση. Τώρα, δέκα χρόνια μετά τη δημοσιονομική κρίση, εγώ είμαι ο τελευταίο που θα σα έλεγε ότι όλα πάνε ρολόι, αλλά ορισμένα θέματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά και αξίζει να το αναφέρουμε. Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και εν μέρη και η Επιτροπή ε, βρίσκονται πίσω από την επιτυχία αυτή. Τώρα είμαστε στο έκτο επακόλουθο ε, έτος ε, ανάπτυξης και στην ε, ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την ε, Ανάπτυξη ε, βλέπουμε ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε ανάπτυξη για έξι συνεχή χρόνια. Όσον αφορά το πληθωρισμό και το λέω προς τους Γερμανούς και Ολλανδούς φίλους που ανησυχούν συνήθως για τον πληθωρισμό είναι στο 1,7%. Μην διαβάζετε λοιπόν μόνο τις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα πράγματα είναι θετικά. Τα ελλείμματα έχουν μειωθεί στο 2,6% από το 6,2% το απόγειο της οικονομικής κρίσης και μόνο μία χώρα και όχι 11 βρίσκονται στη διαδικασία ε, υπερβολικού ελλείμματο. Αυτό δεν σημαίνει την όλα τέλεια. Έχουν γίνει σημαντικέ πρόοδοι όμω και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά τώρα βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν από την κρίση για θέματα ανάπτυξη, απασχόληση και ε, επενδύσεων. Και ε, σχετικά με τις επενδύσεις, αυτό είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Επιτροπή στην αρχή της θητείας της και ο Γενικός Γραμματέας συμμετέσχει ανεργά σε αυτό, δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αυτό που ονομάζουμε και Ταμείο Juncker μερικές φορές και σας ευγνωμονούμε για την υποστήριξή σας. Αυτό αποτελούσε μια επανάσταση στα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έπρεπε να βγάλουμε 60 ε, εκατομμύρια από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να δημιουργήσουμε επενδύσεις. Τέσσερα χρόνια αργότερα μπορούμε να πούμε ότι τώρα βρισκόμαστε στα 400 δισεκατομμύρια τα οποία δημιουργήθηκαν ως επενδύσεις με βάση τα πρώτα, τα πρώτα 60 δισεκατομμύρια που είχαμε χρησιμοποιήσει και αυτό ε, ακολουθείται από ανάπτυξη 1,6% ε, του ΑΕΠ. 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 1,6% ανάπτυξη. Ε, το σχέδιο ποσοτικής χαλάρωσης 2,63 εκατομμύρια και δημιουργεί 1,9% ανάπτυξη. Άρα ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πούμε ότι δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη με πολύ λιγότερα χρήματα, μόνο 400 δισεκατομμύρια σε σχέση με τα 2,6 εκατομμύρια. Επομένω, δεν είναι δίκαιε οι κριτικέ οι οποίε ακούγονται. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι σημαντικό επίτευγμα είναι η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά ε, μέσα σε 20 χρόνια το Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν πέρυσι στο Γκέτεμπουργκ για τις κοινέ αρχές πίσω από τα κοινωνικά δικαιώματα και αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε από κοινού και τα καταφέρνουμε να έχουμε μια κοινή αντίληψη για το ποια είναι αυτά τα πρότυπα. Η κοινή αγορά, η ενιαία αγορά ε, χρειάζεται αυτά τα πρότυπα για να μην υπάρχουν τριβές. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί αυτά τα κοινά πρότυπα ε, την κοινωνική βαθμολογία την οποία καταρτίζει στο πλαίσιο των νέων νομοθετικών μηχανισμών που προτείνονται και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ένα τέταρτο σημείο που θέλω να αναφέρω τώρα είναι το τι κάνουμε σε σχέση με το εμπόριο στην αρχή της θητείας μας ε, και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη τα θέματα του εμπορίου ήταν ιδιαίτερα διχαστικά αλλά αυτό έχει αλλάξει διότι μετά τον Donald Trump και τον Brexit όλοι κατανόησαν ότι όταν υπερασπιζόμαστε ένα διεθνές σύστημα που βασίζεται σε αξίες και κανόνες όταν συνεργαζόμαστε με τους άλλους ε, και ε, εποφελούμαστε όλοι ε, είναι κάτι που είναι προ όφελο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία που καλύπτει το 1 τρίτο του παγκοσμίου ΑΕΠ. Φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο. Έχουμε διδαχθεί και κάτι από το παρελθόν, διότι το εμπόριο φαίνεται να είναι κάτι το αφηρημένο. Και δεν υπάρχουν μόνο νικητέ, αυτό είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν πολλοί νικητέ. Αυτή τη συμφωνία τη διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή σε πλήρη διαφάνεια με το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και έχει φτιάξει και μία ιστοσελίδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με όλε τι λεπτομέρειε ε, για τα αποτελέσματα τη εμπορική αυτή τη συμφωνία για κάθε μία από τι πόλει ε, και τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πάτε στην Ισπανία, και το λέω γιατί ο εισηγητή είναι από την Ισπανία, αλλά θα μπορούσα να σα δώσω παραδείγματα από οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, 6.230 ισπανικέ εταιρείε εξάγουν στην Ιαπωνία το 90% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αν δείτε το χάρτη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής θα δείτε τρεις επιχειρήσεις από τη Σαραγώζα. 41.000 θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν στην Ισπανία από αυτή την εμπορική συμφωνία και συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 740.000 θέσει εργασία. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε στην ιστοσελίδα τη Επιτροπή, να βρείτε τι λεπτομέρειε για την εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία και να πάτε να δείτε ποιο φούρνο ή ποιο χασάπικο στη γειτονιά σα έχει δημιουργήσει θέσει απασχόληση λόγω τη συμφωνία αυτή με την Ιαπωνία. Επομένω, μπορείτε να το πείτε στου πολίτε ότι ε, έχουμε καρπού από τα αποτελέσματα των εργασιών μας και ελπίζω ότι αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για τις ε, εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα άλλο σημείο τώρα για την θητεία του Γενικού Γραμματεία είναι η συμφωνία που επετέχθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου Συμβουλίου και Επιτροπής και τέθηκε σε λειτουργία για τον κανονισμό Προστασία δεδομένων. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνήσαμε για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο με βάση τις κοινέ αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα. Αποφασίσαμε για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι καταρχήν καλό για τους πολίτες, διότι τα δεδομένα τους προστατεύονται καλύτερα. Είναι καλό για τις εταιρείε, διότι υπάρχει μόνο ένα σύστημα κανόνων και όχι 28 διαφορετικά διαφορετικά συστήματα και αυτό δημιουργεί πολλού ε, οι οποίοι μα ακολουθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ιαπωνία έκλεισε αυτή την εμπορική συμφωνία που σα ανέφερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση υιοθέτησε τον δικό μα κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπω και η Βραζιλία και πολλέ χώρε τη Λατινική Αμερική, τμήματα τη Αφρική και εταιρείε όπω η Facebook και η Google υπό την πίεση των σκανδάλων για τα δεδομένα τώρα ε, όλοι ε, διακηρύσουν ότι λατρεύουν τον κανονισμό προσωπικών δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ε, εμείς ε, αποτελούμε το πρότυπο και δεν επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Έχουμε δεσμευθεί ότι σε ένα νέο νομοθετικό κείμενο ότι, που θα τεθεί σε λειτουργία το Δεκέμβριο, ότι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα προστατεύουν τα δεδομένα των πολιτών που έρχονται σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με του θεσμού τη. Έχουμε ένα σημαντικό, σημαντικό ε, σύστημα συμμόρφωση και σα καλούμε να ακολουθήσετε την ίδια πορεία για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων όλων των πολιτών που έρχονται σε επαφή μαζί μας. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή η παρουσίαση που μπορεί να κάνει κανείς για τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής και χάρη και στις ε, αρχές που ασχολούνται με τον προπολογισμό. Επίσης έχουμε επιτύχει πολλά στο παρελθόν. Τώρα τι θα κάνουμε στο μέλλον. Η προετοιμασία των εκλογών και το ποιο θα είναι ο νικητή των εκλογών είναι κάτι το οποίο απασχολεί εσά, του πολιτικού, αλλά και εμά, του διοικητικού τη Επιτροπή, διότι πρέπει να διευκολύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε συμφωνήσει σε μια κοινή διακήρυξη που υπεγράφει από τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρόεδρο Ταγιάννη και τον πρόεδρο του Συμβουλίου και είπαμε ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε για περίπου 100 ακόμη νομοθετικά κείμενα, τα οποία θα πρέπει να είναι έτοιμα πριν τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι, διότι σε μερικά από αυτά τα νομοθετικά κείμενα προχωρούμε γρήγορα, σε άλλα χρειάζεται μεγαλύτερη πρόοδος, διότι οι πολίτες ενδιαφέρονται όχι για μια πρόταση της Επιτροπής, αλλά για κάτι το οποίο είναι γεγονός, έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα και αποτελεί αυτό αποτέλεσμα. Ε, χτες ε, συμφωνήσαμε για τον έλεγχο των ε, άμεσων ξένων επενδύσεων και υπάρχουν υπάρχουν ε, και ευρωβουλευτέ οι οποίοι συμμετέσχουν ενεργά. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γιατί οι ξένε εταιρείε επενδύουν στην Ευρώπη και θέλουμε να δείξουμε ότι έχουμε εργαλεία που προστατεύουν του ε, πολίτε μα ε, και τα συμφέροντά μα. Για πρώτη φορά έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο εργαλείο. Είναι πολύ σημαντικό το ότι παρέχουμε αυτή την προστασία και χρειάζεται πρόοδο και στι υπόλοιπε περίπου 90 νομοθετικέ προτάσει που εκκρεμούν. Εμεί στη Γενική Γραμματεία τη Επιτροπή φροντίζουμε η επόμενη Επιτροπή να είναι σε θέση να αναλάβει τα καθήκοντά της με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ε, και γι' αυτό λαμβάνουμε υπόψη τις συστάσεις της ε, Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και το Σώμα των Επιτρόπων έχει συμφωνήσει για μια μεταρρύθμιση της οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας τελευταία φορά είχε τροποποιηθεί την 1η Ιανουαρίου του 2014. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια λοιπόν μας έχουν δώσει νέα στοιχεία για τις προτεραιότητες, για τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου, για τις σχέσεις ε, με το Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο και για τα θέματα της εξωτερικής διάστασης του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επίση, έχουμε προετοιμάσει μια μεταρρύθμιση τη εταιρική διακυβέρνηση τη Επιτροπή. Ξέρω, κυρία Πρόεδρε και κύριε Σιγητά, αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσά, κύριε Συγήτρια. Έχουμε ένα σύστημα στην Κομισιόν που πιστεύουμε ότι λειτουργεί σωστά, ότι κάθε Γενικό Διευθύντη ε, είναι αρμόδιο για τη διαχείριση στον τομέα του. Αυτοί είναι εξουσιοδοτούντε ε, αξιωματούχοι και αυτό είναι σημαντικό. Το κολέγιο των Επιτρόπων έχει την πολιτική ευθύνη, αλλά τι θα συμβεί αν χρειαστεί κάποιο συντονισμό ε, διυπηρεσιακά. Ε, γι' αυτό το Κολέγιο των Επιτρόπων αύριο το πρωί, αν όλα πάνε καλά, θα υιοθετήσει την επισημοποίηση του ε, Συμβουλίου ε, Εταιρική Διαχείριση, όπω το ονομάζουμε, που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προ το Κολέγιο και θα εκδίδει συστάσει στην υπηρεσία για οριζόντια θέματα, κυρίω για την ασφάλεια πληροφορική, για την καλύτερη προετοιμασία μα σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο ως επίσης και για την υλοποίηση των νόμων προστασίας δεδομένων στην Κομισιόν και για την παρακολούθηση των δύο συστάσεων της Όλαφ. Έχουμε μια δομή σε κάθε σύσταση της Όλαφ για να αποφεύγουμε την απάτη ε, συστημικά να υπάρχει και ένα οργάνο που θα το συνιστά αυτό ε, και θα το υλοποιεί χωρίς ε, να αμφισβητείται η αρμοδιότητα των επιμέρους Γενικών Διευθυντών και του Κολεγίου των Επιτρόπων. Αυτή η μεταρρύθμιση θα υιοθετηθεί αύριο όλα πάνε καλά και θα είναι μια πλήρης υλοποίηση όλων των συστάσεων. Ε, μεταρρυθμίζουμε την συνεργασία μας με την Όλαφ. Υπήρξε κάποια επιφύλαξη για το πώς λειτουργούσε το παρελθόν εδώ πέρα. Θα έχουμε τον νέο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ ε, που τον έχετε συναντήσει ήδη και αφού έχουμε και νέο Γενικό Γραμματέα συμφωνήσαμε μια νέα μορφή συνεργασίας ώστε οι ερευνητικές δυνατότητες της Όλαφ να παραμείνουν αυτόνομες και ανεξάρτητες και έτσι καταργούμε τον οικό εκαθάριση του clearing house που κάποιοι από εσά επέκριναν γιατί πιστεύω ότι δεν το χρειαζόμαστε πλέον. Όταν θα υπάρξει σύσταση πολιτική από την Όλαφ, το ε, Συμβούλιο Διακυβέρνηση τη Κομισιόν θα φροντίζει όλε τι συστάσει τη Όλαφ να υλοποιούνται σε όλη την Κομισιόν. Μίλησα λίγο περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν, κυρίε και κύριοι, αλλά επειδή ήταν η πρώτη φορά, θέλησα να σα τα πω ε, εκτενώς και να με γνωρίσετε και καλύτερα. Πιστεύω ότι ναι, πολλά είναι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές είναι προκλήσεις και το Brexit βλέπουμε αυτή τη βδομάδα, πρέπει να φτάσει στο τέλος του, να οριστικοποιηθεί. Πολλοί κόσμος δουλεύει στην Κομισιόν γι' αυτό και ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι αν θα καταφέρουμε να έχουμε μια συμφωνία την Κυριακή. Έχουμε και άλλες προκλήσεις στο κράτος δικαίου, τη δημοσιονομική κατάσταση σε ορισμένα κρατημέλη, το λαϊκισμό σε πολλές χώρες, αλλά κάποια φορά πρέπει να καθόμαστε και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και επιτυχίε, Υπάρχουν και πρόοδοι. Δεν είναι όλα τέλεια. Ποτέ δεν θα είναι όλα τέλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μερικέ φορέ θα πρέπει να δείχνουμε λίγο μεγαλύτερη περηφάνεια για το όσο έχουμε επιτύχει χάρη στη δουλειά του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και λίγο τη Επιτροπή. Παρότι φυσικά είμαστε λιγότερο σημαντικοί σε αυτό το, σε αυτό το τρίγωνο θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ πολύ και αναμένω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε κατευθείαν στη συζήτηση. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας κύριε Ρούσο. Θα σας δώσουμε το λόγο για να κάνετε την εισαγωγή στο κεφάλαιο. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που καθυστέρησα. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Εισηγήτρια, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του Ελέγχου του Προϋπολογισμού, είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο 10 του ελεκτικού συνεδρίου της ε, έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για την αξιολόγηση των διοικητικών δαπανών, ε, συγκεκριμένα της Επιτροπής. Η αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου για την ετήσια έκθεση του 2017 είναι θετική. Οι διοικητικές δαπάνες δεν επηρεάζονται από σφάλμα σημαντικότητας. Έχουμε εντοπίσει ποσοστό σφάλματος κατεκτήμηση 0,5%. Η αξιολόγηση βασίζεται σε δείγμα 55 συναλλαγών, εκ των οποίων 26 σχετίζονταν με την Κομισιόν. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώσαμε μικρό αριθμό σφαλμάτων σε σχέση με δαπάνες προσωπικού και κάποιες αδυναμίες στην διαχείριση PMO των οικογενειακών επιδομάτων. Τα εξετάζουμε εκτενώς με τη διοίκηση της Κομισιόν. Αυτά είναι τα ευρήματα του ελέγχου μας για το έτος 2017. Σας ε, προτείνουμε λοιπόν η Κομισιόν να βελτιώσει το, το σύστημά της διαχείρισης των νόμιμων οικογενειακών επιδομάτων με διαρκής ελέγχους ε, συμμόρφωσης ε, για τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνουν τα μέλη του προσωπικού από άλλες πηγές. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια, κυρία Γιάλα Ζέντερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ρούσο, που ήταν πολύ σύντομος. Και θα ήθελα βεβαίως να ε, ευχηθώ καλώς όρισε στον κύριο Σελμάιερ που όπως είπε και η πρόεδρος μας τόσες φορές τον αναφέραμε την απουσία του και πια έχουμε τη δυνατότητα ε, να τον συναντήσουμε και μπορούμε να του υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις και να ρωτήσουμε και αυτά που θα ρωτούσαν οι συνάδελφοι αν ήταν εδώ. Να σας πω καταρχήν πως πρέπει να επαναλάβω το εξής. Η παρουσίαση που μας κάνατε, τουλάχιστον για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, που είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε, στην πρόταση την οποία θα υποβάλλουμε στη διάρκεια της ε, διαδικασίας απαλλαγής είναι μία παρουσίαση καλή. Αλλά σε καθημερινό επίπεδο πρέπει να σας πω πως το 2016, όχι το 2013, το 2016 έγινε το δημοψήφισμα για το Brexit, ένα θέμα το οποίο ακόμα, για το οποίο ακόμα θα ακούσει θα κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Σε ευχαριστώ που το ανέφερες και αυτή τη στιγμή έχουμε για παράδειγμα καλές εταιρείες από τη Σαραγώσα που έχουν ευκαιρίες στην Ιαπωνία αλλά Σκεφτείτε πόσε είναι οι εταιρείε τη Ισπανία που κάνουν εξαγωγέ στην Ισπανία. Πόσοι Βρετανοί υπήκοοι ζουν στην Ισπανία. Και αυτή τη στιγμή παίρνουν δύσκολε στιγμέ. Και τι συμβαίνει με όλου του Ισπανού που μετανάστευσαν ε, ε, στην ε, Βρετανία λόγω τη κρίση το 2008 και που αναρωτιούνται αύριο τι θα του συμβεί. Οπότε σα ευχαριστώ πολύ που το αναφέρατε γιατί θα χρησιμοποιήσω και τα παραδείγματα που βάλατε και καλό είναι στις περιπτώσεις που έχουμε θετικά μηνύματα να το λέμε, να το αναγνωρίζουμε, να μην το λένε μόνο οι τρίτες χώρες, αλλά και εμείς να αναγνωρίσουμε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να γνωρούμε πως σήμερα είμαστε σε μια κατάσταση όπου καλό θα ήταν να δώσουμε κάποιες εξηγήσει για τα όσα μας συμβαίνουν. Και είναι σημαντικό που ο Γενικό Γραμματέα, γιατί εγώ με τον κύριο Ιταλιάνερ δεν τα πήγαινα καλά καθόλου, και ούτε απαντούσε καν σε αυτά που του έλεγα. Νομίζω δεν με άκουγε καν και εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος όταν τα πάνε καλά μαζί μου. Όταν δεν τα πάνε καλά μαζί μου, δεν θα πω κάτι το οποίο είναι χιδαίο γιατί θα με μεταφράσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει η στάση μου είναι αρνητική. Εσείς είστε γενικός γραμματέας και μετά θα μιλήσουμε για τους διορισμούς. Ως γενικός γραμματέας ελπίζω πώς θα τα πάτε καλύτερα μαζί μου και εγώ μαζί σας. Γιατί για κάποιες από τις απαντήσεις που δώσατε, για παράδειγμα κυβερνοασφάλεια, δεν είναι δική σα ευθύνη, αλλά εσείς κάνετε ό,τι μπορείτε για να λειτουργήσουν τα κράτη-μέλη, σας ευχαριστώ, αλλά για άλλα θέματα και απαντήσεις που έχουν να κάνουν με τις διαδικασίες, τις εσωτερικές, το κομμάτι που είναι συντονισμός, εναρμόνιση, όπως επίσης και οι διορισμοί, οι οποίοι όντως επηρεάζουν την καλή φήμη των θεσμών, ε, εκεί οι απαντήσεις το λέω με κάθε καλή διάθεση, ε, ήταν λίγο υπερβολικές. Και το λέμε έτσι στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γιατί όταν μιλάμε για απαντήσεις στις δικές μας ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω πως οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι πολύ πιο επαγγελματικές. Και όχι τσαπατσούλικες. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια εσεί θεωρείτε πως σε κάποιους διορισμού και δεν το προσωποποιώ. Μιλώ για γενικούς διευθυντέ και Για τον κύριο Ιταλιάνερα α πούμε έχω πει πολλά. Ήταν μια σειρά από διορισμού, οι οποίοι επηρεάζουν το πώς μας βλέπουν τη φήμη των ε, θεσμών, όσο μη και να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και όπου μας συζήτησαν και στον τύπο και εντός ε, και εκτό ε, θεσμών και όπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργήθηκε μια κατάσταση, για να το πω έτσι ευγενικά, ταραχώδη. Τα σημαντικά λοιπόν σημεία θα πρέπει να είναι στο θεματολόγιο ε, του, ε, των επιτρόπων. Ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα δεν είναι ένα μικρό θέμα. Σίγουρα πρέπει να περάσει από τους επιτρόπους. Και θα πρέπει όμως να γίνεται με διάφανο τρόπο για όλο το συλλογικό όργανο των επιτρόπων. Διαφορετικά θα πιστέψουμε κι εμείς πως υπάρχει πρόβλημα. Και όταν μου λέτε στις απαντήσεις σας πως η ισορροπία μεταξύ φύλων είναι καλύτερη αν γίνει ε, μέσω μεταφοράς, να μου το εξηγήσετε. Γιατί δεν καταλαβαίνω πως σε μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά χειραγωγείται ε, και τους υποδεικνύουμε με το δάχτυλο, τότε δεν καταλαβαίνω τι ε, τι ε, κίνητρα δίνουμε στις γυναίκες υπαλλήλους για να καταθέσουν υποψηφιότητες. Εντάξει, όταν μιλάμε για γενικό διευθυντή, για ε, υποδιευθυντή και τέτοιου είδους θέσει, θα πρέπει η κατάσταση να είναι πιο διάφανη και η ισορροπία μεταξύ φύλων δεν θα πρέπει να γίνεται και να είναι γυναίκες δακτυλοδεικτούμενες, αλλά θα πρέπει να γίνεται μια προηγούμενη, σε μια προηγούμενη φάση όπου θα ενθαρρύνουμε τις γυναίκες υπαλλήλου να καταθέτουν υποψηφιότητα και όχι να τις αποτρέπουμε καθόλου αυτή τη διαδικασία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Στι επόμενε λοιπόν απαντήσει, τι οποίε σίγουρα θα χρειαστεί να μου στείλετε και στην οποία θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε μέχρι να κατατεθεί η ε, εκθέση, καλό θα είναι όλα αυτά να τα βελτιώσουμε. για τον τρόπο που διαχειρίζετε εσεί τα θέματα ω γενικό Γραμματέας. Συντονισμός και εναρμόνιση μεθοδολογία των Γενικών Διευθύνσεων. Και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω αύριο να μα παρουσιάσει όταν εγκριθεί το έγγραφο για τον συντονισμό Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να έχουμε ιδιωτικά στελέχη που διορίζονται στο δημόσιο, γιατί συνήθως γίνεται σε κρίσιμες στιγμές, αλλά αυτό η ονομασία του Διοικητικού Συμβούλου, του εταιρική, ε, Εταιρικό Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι όπως το έχετε ονομάσει, εν πάση περιπτώσει δεν με ικανοποιεί, αλλά αν είναι να βελτιώσει την κατάσταση σε επίπεδο συντονισμού και εναρμόνισης, εντάξει. Γιατί εγώ είχα μεγάλα προβλήματα για τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται μεταξύ τους οι γενικές διευθύνσεις. Και όταν κοιτά κανείς τα αποτελέσματα, ξεκάθαρα τα και αποκλειστικά και μόνο τα αποτελέσματα. Θα δείτε ότι στη Γενική Διεύθυνση ταξούντ ακολουθούν μια πολιτική και όταν έχουμε πολιτική, ε, ε, εξωτερική πολιτική ε, είναι τελείως διαφορετική. Γιατί κάνετε, συσφίγγετε σχέσεις σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων και μετά έρχεται η κυρία Γιούροβα και δίνει ένα χαστούκι γιατί υπάρχουν κάποια θέματα ανταγωνισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός έγκυρης προειδοποίησης για να μην πέφτουμε σε τέτοιου είδους αντιφάσεις, γιατί αυτό πλήττει και τη φήμη μας. Εναρμόνιση μεθοδολογίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Πρώτη φορά είστε εσείς εδώ, αλλά στι διάφορε ακροασει που έγιναν στι επιτροπέ και στι γενικέ διευθύνσει. είδαμε πω ένα θέμα τόσο σημαντικό που είναι η μέτρηση του ποσοστού σφάλματο στην εσωτερικό έλεγχο όπου χρειάζεται να ειδοποιήσουμε το ποσοστό σφάλματος. Έχουμε το εναπομείνον ε, ποσοστό σφάλματος και αυτό θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τελικά κάθε <laughs> γενική διεύθυνση έχει το δικό της τρόπο που το υπολογίζει. Άλλα κάνει DG Agri, άλλοι κάνει DG ε, Deve κτλ. Ο καθένας δηλαδή ακολουθεί τη δική του μέθοδο. για αυτό το υπολοιπόμενο ποσοστό σφάλματος που δυσκολεύει την κατάσταση και που κάνει πολύ δύσκολη την προσπάθεια σύγκρισης. Γιατί βέβαια χρειάζεται να βλέπουμε ποιος πάει πιο καλά και ποιος χειρότερα. Και ουσιαστικά αυτό μας οδηγεί σε κάποιες αντιφάσεις τη στιγμή ε, της συνεργασίας μας με το ελεγκτικό συνέδριο. Και αυτά είναι σημαντικά σημεία που θα πρέπει να τα δείτε και τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια στα πλαίσια της ε, ε, τρέχουσας διαδικασίας απαλλαγής. Τα λέω αυτά γιατί μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο θα πρέπει και εμείς να μπορούμε να αποφασίσουμε πώς μετράμε το κομμάτι που είναι λογιστικό και το κομμάτι το οποίο είναι εσωτερικού ελέγχου για να μπορούμε να τα συγκρίνουμε και πώς μπορούμε να συγκρίνουμε μεταξύ τους και τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα. Στη διαδικασία αυτή που έχουμε την ακρόαση του ελεγκτικού συνεδρίου, έχω κάποιες αμφιβολίες. Ε, χαίρομαι που μας εξηγήσατε ε, ε ποιος, ποια είναι η εντολή του Γενικού Γραμματέα. Πολλές φορές από πρόεδρο σε πρόεδρο αυτό αλλάζει, αλλά ε, για την διαδικασία, την καταντιμολία που έχουμε με το ελεγκτικό συνέδριο, θα ήθελα να μου εξηγήσετε με ποιο τρόπο εσείς θα καταφέρετε αυτή η διαδικασία να είναι επαρκώς διάφανη και επαγγελματική. Να δείχνει λοιπόν επαγγελματισμό για να μην έχουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας την εντύπωση πως τα συμπεράσματα οδηγούν σε ότι βελτιώνονται τα πράγματα χωρίς να διορθώνονται. Ότι βελτιώνονται εντάξει, αλλά χρειάζεται και να διορθωθούν. Αυτή είναι η προσωπική μου μάχη. Γιατί αν απλώς φτιασιδώνονται, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Θα θέλαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με έναν τρόπο πιο επαγγελματικό. Αυτό να κάνετε στη νέα εντολή που έχετε. Να αντιμετωπίσετε τα θέματα και να τα βελτιώνετε. Και εγώ θα είμαι η πρώτη που θα σας στηρίξω. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα για τα υπόλοιπα. Μήπως οι συνάδελφοι θέλουν να πούν το λόγο. Μετά μπορώ να ξαναμιλήσω. Πείτε Παρακαλώ, κύριε Σελμάγερ. Ευχαριστώ, κύριε Συγητρία, κύριε Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Να απαντήσω με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις. Επανέρχομαι και σε αυτό που είπε ο εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου για το ένα σημείο ότι παρότι δεν έχουμε ε, ουσιαστικό σφάλμα. Είπε ότι υπήρχαν κάποιες αδυναμίε στο πώς έγινε η διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων. Το αναγνωρίζουμε αυτό και η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για βελτίωση. Έχει ένα σύστημα παρακολούθησης ούτω ώστε το προσωπικό να δηλώνει ετησίω τα οικογενειακά επιδόματα που λαμβάνει από άλλε πηγέ εκτό Επιτροπή με ένα ειδικό σύστημα πληροφορικής αυτό ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπίσει το ζήτημα που είχαμε. Επίσης, κάποια επιδόματα που δόθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα ε, ε, οδήγησε στο να κάνουμε επικαιροποιήσει σε ε, μικρά χρονικά διαστήματα για να καλύψουμε και αυτές τις δυνατότητες και η έλεγχή μα να είναι περισσότερο αποτελεσματική. Επίσης, κάνουμε ανακοινώσει προ το προσωπικό βελτιώνοντας την επίγνωση του προσωπικού για τα θέματα αυτά ούτως ώστε να ενημερώνονται οι φάκελοι αυτόματα. Συμφωνούμε λοιπόν με τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ήδη υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης. Ευχαριστούμε λοιπόν το Συμβούλιο, το, το Ελεγκτικό Συνέδριο που είδαν ότι δεν υπήρχε και περιθώριο ε, ουσιαστικού σφάλματος. Προς την κυρία Γιάλα, καταρχήν συμμερίζομαι με τις ανησυχίες σας για την αβεβαιότητα που δημιουργεί το Brexit. Παρ' όλα αυτά κάνω έκκληση προς όλους σας, ε, ε, λέγοντάς σας ότι δεν το δημιουργήσαμε εμείς το Brexit, το δημιουργήσε το Ηνωμένο Βασίλειο με την απόφασή του, την σεβόμαστε. Μας θλίβει αλλά δεν ε, δημιουργήσαμε εμείς το χάος αυτό. Εμείς διαπραγματευθήκαμε επαγγελματικά επί δύο χρόνια, έχουμε μια πολύ καλή διαδικασία, ένα πολύ καλό διαπραγματευτή και τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το Ηνωμένο ε, Βασίλειο συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όταν είμαστε ενωμένοι προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, είτε στο Brexit, έναντι του Πρόεδρου Τραμπ, πάντοτε το να είμαστε ενωμένοι με μια φωνή, αυτό είναι θετικό. Ελπίζουμε να συμφωνηθεί συζητηθούν ε, τα αντικείμενα τη διαπραγματεύση και να επικυρωθούν, που είναι ένα άλλο θέμα η επικύρωση. Σα ευχαριστούμε για την ενθάρρυνσή σα μα έχουν ενθαρρύνει και τα κρατημέλη και στην ε, Γενική Γραμματεία τη Επιτροπή. Έχουμε μια task force για την ετοιμότητα σε θέματα Brexit. Αυτή η task force είναι μια μονάδα που προετοιμάζεται για τι συνέπειε του Brexit. Είναι πραγματικά ε, θλιβερό το, το έργο του και του επισκέπτομαι συχνά και του ενθαρρύνω γιατί ασχολούνται με το απεσιόδοξο σενάριο. Τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική θέση του ε, κ. Μπαχνιέ, ε, διότι θέλουμε να έχουμε διαπραγμάτευση, αλλά θέλουμε να δούμε ε, πώ θα είμαστε προετοιμασμένοι και για οτιδήποτε αρνητικό. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι και αν συμβεί, κάποια θέματα που θα είναι το αποτέλεσμα του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει τρίτη χώρα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο νομικό πλαίσιο. Τι θα γίνει με του κανονισμού για τη θεώρηση διαβατηρίου, τι θα γίνει για του στόχου αποτελεσματικότητα που είχαν συμφωνηθεί για τα 28 κράτη-μέλη και τώρα θα πρέπει να συμφωνηθούν εκ νέου για τα 27. Τι θα γίνει με τους οργανισμούς που είχαν έδρα το Λονδίνο. Έχουμε συμφωνήσει για την μετακίνησή του για την αρχή των φαρμάκων που δεν είναι ένας οργανισμός με γραφειοκράτες απλώς, είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για τη δημόσια υγεία και για την ενιαία αγορά. Και αν περιμέναμε περισσότερο μέχρι να το κάνουμε αυτό, όλοι αυτοί οι πολίτες, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι δεν θα είχαν κανένα λόγο να μείνουν στον οργανισμό. Θα είχαμε χάσει όλους τους εμπειρογνώμονες, όλα τα ταλέντα που έχουμε συγκεντρώσει σε αυτόν τον οργανισμό. Ευχαριστώ λοιπόν και το Κοινοβούλιο που μας έχει βοηθήσει να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε για πάνω από χίλια άτομα, ώστε να προσπαθήσουμε να τους κρατήσουμε στον οργανισμό παρά τη μετακίνηση που δημιουργεί προβλήματα για τους ίδιους και τι οικογένειε. τους. Συμφωνώ με την κυρία Γιάλα όταν λέει ότι πρέπει να τονίζουμε τα θετικά χωρί να υποτιμούμε τις δυσκολίες επειδή μιλήσατε και για τον προκάτοχό μου με σκληρά λόγια, ε, εγώ δεν μιλώ ποτέ για κάποιον που δεν είναι παρόν στην αίθουσα, οπότε δεν θα πω κουβέντα για τους προκατόχους μου, αλλά δεν ε, είναι ίδιόν μου να μιλώ για τους προκατόχους. Ε, αν υπάρχουν επικρίσεις, παρακαλώ να καλέσετε τους προκατόχους μου και να τα συζητήσετε μαζί τους. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα για τον προκατοχό μου και φαντάζομαι ότι κατανοείτε τη θέση μου. Για το, τα πιο γενικά θέματα που αναφέρατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα αυτά, για το θέμα της ισότητας των φύλων. Ελπίζω ότι το γνωρίζετε, κυρία Γιάλα. Αν δεν το γνωρίζετε, πρέπει να το πω εγώ εδώ ότι από τότε που είμαι στην Επιτροπή και σε μία ε, θέση ε, προϊσταμένου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, Πάντοτε προσπαθώ να μιλήσω για ποσοστώσεις σχετικά με γυναικείες θέσεις απασχόλησης στην Επιτροπή και όχι μόνο στην Επιτροπή. Και έχω ζητήσει και το να συνταχθεί μια πρόταση για ποσοστώσει σε διοικητικά συμβούλια εταιριών. Και αυτή η Επιτροπή με τον πρόεδρο Γιούνκερ, με την κυρία Γεωργίευα τότε και τον κύριο Έτιγκερ τώρα, ακολουθεί μια πολιτική τουλάχιστον 40% ποσόστοση τις ανώτερε ε, θέσει, ανώτερες και μέσες διοικητικές θέσει και έχουμε κάνει εξαιρετική πρόοδο. Δεν ήταν καθόλου εύκολο και δεν έχει καταφέρει να το κάνει ούτε η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ούτε τα κράτη-μέλη. Όμω στη Γενική Γραμματεία το έχουμε καταφέρει από τότε που είμαι εγώ επικεφαλή. Έχουμε βελτιώσει κατά 10% τον αριθμό των γυναικών στελεχών. Δεν τα έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Υπάρχει και ένα πρόγραμμα ανάπτυξη γυναικείων ταλέντων στην Επιτροπή και πρέπει να ενθαρρύνουμε τι γυναίκε. Εάν δείτε τις ε, τρεις ε, ε, τις ε, τρεις βοηθούς μου, τις τρεις αναπληρώτριές μου είναι τρεις γυναίκες. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν γιατί έχω τρεις γυναίκες αναπληρώτριες στη θέση του Γενικού Γραμματέα δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να φτάσουμε εκεί που θέλουμε και μια και δεν είμαστε στο 1918 αλλά στο 2018 θα έπρεπε τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ικανοποιημένοι από την παρούσα κατάσταση. Αλλά ελπίζω ότι σύντομα θα πούμε ότι έχουμε επιτύχει του στόχου μα και προωθούμε το ταλέντο μεταξύ των γυναικών και όχι μόνο μεταξύ των γυναικών αλλά και ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών για να υπάρχει ισότητα. Και αυτό διότι πιστεύουμε και εγώ προσωπικά ως μάνατζερ πιστεύω ότι η διαφοροποίηση μέσα στις ομάδες είναι θετικό. Η ομάδα δουλεύει καλύτερα γιατί ε, όταν έχουμε ε, διαφορετικά φύλλα, διαφορετικές εθνικότητες ε, και διαφορετικά υπόβαθρα, πάντοτε η ομαδική δουλειά γίνεται καλύτερη. Κάνετε ερωτήσεις και για το διορισμό μου. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπορώ να σας πω πολλά από αυτού γιατί εγώ δεν ήμουν τμήμα της διαδικασίας διορισμού μου, ήμουν το αντικείμενο αντικείμενο του διορισμού και χαίρομαι για την ομόφωνη ε, έγκριση που με έδωσε το ε, Σώμα των Επιτρόπων και είμαι ε, υπερήφανος για τις υπηρεσίες μου, τις οποίες δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς από εσά. Έχουν λεχθεί πολλά, αλλά ποτέ δεν μου έχουν πει κάτι πολύ συγκεκριμένο για την όλη διαδικασία. Νομίζω ότι όλα ήταν βάση των κανόνων. Το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε τις κατάλληλες αποφάσεις και ελπίζω ότι θα είστε κι εσείς ε, σίγουροι ότι η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με τους προκατόχους μου. Δεν ξέρω γιατί επικεντρώνεται η προσοχή στο δικό μου πρόσωπο και όχι στους προηγούμενους. Ίσως να έχει σχέση με το Brexit, ίσως να έχει σχέση με άλλες διαδικασίες. Μπορείτε να με επικρίνετε για τις προσωπικές μου επιλογές, αλλά ε, όχι για τις διαδικασίες οι οποίες ήταν απόλυτα νόμιμες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, διότι δεν ήμουν στην αίθουσα. Όπως ε, γίνεται πάντοτε, δεν συμμετέχουν ε, οι ίδιοι ε, ε, οι προϊστάμενοι όταν ε, εκλέγονται στη διαδικασία επιλογής τους. Τώρα, για αυτό το Συμβούλιο εταιρική Διαχείρισης θέλω να πω ότι ο ρόλος του είναι να εξετάζει θέματα που είναι αρμοδιότητες της κάθε Γενικής Διεύθυνσης στην καθημερινή της δουλειά δεν είναι πολιτικό σώμα. Εμείς κάνουμε μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ της ε, διοικητικής ε, καθημερινότητας και της πολιτικής διαχείρισης από τους επιτρόπους. Έχουμε και μια πολιτική επιτροπή ως έννοια την οποία έχει προκηρύξει ο πρόεδρος Γιούγκερ, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Όλες οι πολιτικές αποφάσεις λαμβάνουν οι επιτροποί. Οπότε αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των απόψεων ε, Γιούροβα και Μοσκοβισή, αυτό θα συζητηθεί από τους επιτρόπους ανθρώπους στο συλλογικό όργανο των επιτρόπων. Αν υπάρχει θέμα διαχειριστικό, δηλαδή απόκληση στα ποσοστά ασφάλματος, ναι, τότε όντως θα είναι η Γενική Διεύθυνση ε, που θα το συζητήσει. Και επίσης αυτό το Εταιρικό Διοικητικό Συμβούλιο για το οποίο εγώ είμαι αρμόδιος. Θα είμαι μάλλον, γιατί ακόμα δεν μου έχει αποδοθεί αυτή η αρμοδιότητα. Τώρα για την ε, δομή που έχει δώσει ο πρόεδρος Γιούνκερ ε, σε αυτή την επιτροπή να σας πω πως καταρχήν δεν έχει αλλάξει ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα. Από τον Εμμανουέλ Στάιν το ίδιο είναι. Η περιγραφή των καθηκόντων και οι τρεις λειτουργίες που έχουμε είναι αυτά τα οποία σας περιέγραψα, δεν έχουν αλλάξει καθόλου και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση αλλαγής. Όμως, για τη δομή ε, με τις, με τις αντιπροεδρίες που ε, εισήγαγε ο πρόεδρος Γιούγκερ ε, οδήγησε στο εξή να μην έχουμε αντιφατικές πρωτοβουλίες από τις διάφορες υπηρεσίες και αυτό είναι και το ποθητό αποτέλεσμα. Στο παρελθόν είχαμε στην χάραξη πολιτικής μια πολιτική bottom-up το οποίο σημαίνει ότι είχαμε πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν ήταν συντονισμένες μεταξύ τους. Σήμερα έχουμε την αντίστροφη διαδικασία. Ο πρόεδρος που είναι υποψήφιος πηγαίνει στο κοινοβούλιο και κάνει ενό είδου πολιτικής συμφωνίας. Ε, το έκανε το 2014. Αυτές είναι 10 προτεραιότητες, τι οποίε θα παραδώσω και αυτές εφαρμόζονται από τις αντιπροεδρίες μέσω κάποιων ομάδων project team από του επιτρόπου. Οπότε περνά από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Πετροπή. εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο πολλές φορές, ε, εφαρμόστηκαν από το, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, οδήγησε σε, ένα 25, μια μείωση 25% ε, του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί τότε συμφωνήσατε με τον κύριο Γιούνκερ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει λιγότερο και πιο αποτελεσματικά. Το κάναμε. Το είχε πει και το ελεγκτικό συνέδριο δεν ήταν δική μου επιλογή και οδήγησε στο εξή αποτέλεσμα να είναι υπό περισσότερη καθοδήγηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να είναι αρμόδιο για όλες τι επιλογές του όργανο των επιτρόπων. Άλλο ένα παράδειγμα είναι οι πρωτοβουλίε των πολιτών, που ξέρω ότι για πολλού είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Στην προηγούμενη θητεία τη Επιτροπή. ο Γενικό Γραμματείας αναλάμβανε να χειριστεί αυτέ τι πρωτοβουλίε πολιτών. Δηλαδή θα ερχόταν κάτι, μια πρωτοβουλία κατά της TTIP, της συμφωνίας αυτής. Το κατά πόσο είναι παραδεκτό, που είναι νομική βάση στα πλαίσια του κανονισμού, ε, ήταν μια απόφαση που ελάμβανε σε συμφωνία με τη νομική υπηρεσία η Γενική Γραμματεία. Όταν έγινε πρόεδρος ο, πρόεδρος Γιούγκερ ρώτησε του επιτρόπου από την προηγούμενη ε, επιτροπή και είπε τι, θα αλλάξει, τι θέλετε να αλλάξετε και είπε, είπανε ότι θέλουμε επειδή είναι πολύ σημαντικό ε, να αποφασίζουμε στο συλλογικό όργανο των επιτρόπων τι θα γίνεται με τις πρωτοβουλίες πολιτών γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ε, αυτό έγινε και γίνεται μια προφορική συζήτηση σε επίπεδο ε, συλλογικό οργάνου των ε, ε, επιτρόπων. Και γι' αυτό είναι πιο φιλικές προς τον πολίτη οι πρωτοβουλίες των πολιτών σήμερα. Και αν δεν είναι εξαιρετικά διατυπωμένοι αλλά για παράδειγμα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι παραδεκτό, τότε θα Κρυθεί, μερικώς ε, παραδεκτή η πρωτοβουλία αυτή και κάθε δύο εβδομάδες στέλνουμε και το ανακοινωθέν τύπου έτσι ώστε να φαίνεται ότι αυτά έχουν συζητηθεί από τους ε, πολίτες ότι οι πρωτοβουλίες είναι εκεί και δεν είναι κάτι το οποίο έχει αφαιθεί στη διοίκηση να αποφασίζει, αλλά αποφασίζει από επιτρόπου οι οποίοι λογοδοτούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Γιάλα, για το θέμα του ποσοστού σφάλματο, το μόνο που μπορώ να σα πω είναι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το σύστημα να είναι το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Έχω μόλι υπογράψει μια επιστολή προ όλε τι γενικέ διευθύνσει, έτσι ώστε για την επόμενη χρονιά, όπου θα είμαι υπεύθυνο, εσεί μιλάτε για το 17, εγώ δεν ήμουν ε, διορισμένος τότε, για φέτος είμαι και το υπέγραψα μόλις για να είμαστε σίγουροι πως θα είμαστε όσο το δυνατόν πιο συνεκτικοί και μπαίνοντα στι λεπτομέρειε στο θέμα των ε, ποσοστών ε, σφάλματο και του υπολοιπόμενου ποσοστού σφάλματο, είναι περίπλοκο το θέμα. Έχει να κάνει με, την πολυετή φύση του προπολογισμού μα. Υπάρχουν διαφορετικέ εκτιμήσει μεταξύ ημών ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και ημών με ύψιλον αλλά θέλω να δείτε τι έχουν κάνει οι προκατοχοί μου. Κάναν ό,τι μπορούσαν. Αν με στηρίξετε περισσότερο, θα προσπαθήσω να τα πάω ακόμα καλύτερα. Σα ευχαριστώ πολύ και προσδοκώ και με εσά, κυρία Γιάλα, στενή συνεργασία και σα ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σα λόγια. Πραγματικά το εκτιμώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σκιώδη συζητητέ. Ξεκινώ με το ΕΛΚ και με τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τι ενημερώσει αυτέ και πρέπει να πούμε και για τα πρακτικά ότι ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα είναι θέμα διαφορετικής απόφασης. Αύριο θα το συζητήσουμε και με την Επιτροπή ε, Αναφορών όταν θα συζητήσουμε το σχετικό θέμα. Εμείς χαιρόμαστε να σας έχουμε ε, στο πλευρό μας διότι είναι αποδεδειγμένο ότι μπορείτε να προσφέρετε. Το πρώτο το οποίο αναφέρεται είναι το τέλος της διαδικασίας του Clearing House, το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό για την ανεξαρτησία της Όλαφ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ένα δεύτερο θέμα που αναφέρεται, το Corporate Management Board, είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αύριο στο Σώμα των Επιτρόπων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στο σχετικό κείμενο, γιατί θέλουμε να το εξετάσουμε. Ένα άλλο σημείο ε, ο εσωτερικό έλεγχο εξέτασε ορισμένα θέματα που μα είναι πολύ ενδιαφέροντα και εμεί ω Ευρωβουλευτέ θέλουμε να τα εξετάσουμε. Το θέμα, το τι γίνεται με τι γραπτέ ερωτήσει των Ευρωβουλευτών. Έχετε τι κοινοβουλευτικέ ερωτήσει ω αρμοδιότητα. Ε, ίσως ο εσωτερικός έλεγχος δεν γράφει μεγάλα κείμενα, παρακαλούμε, όταν υπάρχει μια μεγάλη διοικητική διαδικασία ε, τουλάχιστον ε, οι απαντήσεις να αξίζουν το χαρτί στο οποίο είναι γραμμένες ε, και οι γραπτές ερωτήσεις των συναδέλφων να μπορούν να απαντώνται κατά τρόπο που θα είναι αντίστοιχος στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου. Ένα δεύτερο σημείο σχετικά με τη διακυβέρνηση. Στην έκθεση εσωτερικού ελέγχου το έχουμε αναφέρει. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων που δεν προετοιμάζονται από την Eurostat. Τις έχουμε διατυπώσει αυτές τις αμφιβολίες μας εδώ και πολύ καιρό. Θα θέλαμε να έχουμε μια επιβεβαίωση για τι στατιστικά στοιχεία μιλάμε. Καλό θα ήταν αν είχατε να προσθέσετε κάτι γι' αυτό. η αλλαγή για ε, την Επιτροπή ε, Audit Progress ε, είναι κάτι στο οποίο καλό θα ήταν να μας δίνετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς κάνουν οι επίτροποι για τη διαχείριση, την εσωτερική διαχείριση. Ένα τρίτο σημείο αφορά τις περικοπές προσωπικού. Ε, υπάρχουν περικοπές σε σχέση με το 2013. Ε, δημιουργήθηκε μια νέα κατηγορία, μειώθηκε η κατηγορία D και αυξήθηκε η κατηγορία AS. Αυξήθηκαν ε, οι συμβασιούχοι. Πάντως υπάρχει μια σημαντική αύξηση από το 2013. θα μπορούσαμε να έχουμε μια εξοικονόμηση θέσεων. Ε, σήμερα υπάρχουν λιγότερες ε, ε, υπερορίες που δεν καλύπτονται σε σχέση με παλαιότερα, οπότε δεν ξέρω αυτό πώς μπορούμε να το σχολιάσουμε. Ε, υπάρχουν ορισμένα σημεία στα οποία παρακάμπτεται ο κανονισμός ε, του προσωπικού. Έχουμε 65 από το 2017, 9 συμβούλου. Πώς βλέπετε το σύστημα των προαγωγών και ε, αυτή της παράκαμψης των διατάξεων. Και για το EPSC θα ήθελα να μας πείτε κάτι παραπάνω. Θα δώσω όμως ε, τώρα το λόγο στους άλλους και τον κύριο Γκεμπράντη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα που βρίσκεστε εδώ ανάμεσά μας. Δεν θα είμαι πολύ επικριτικός γιατί είναι η πρώτη σας φορά εδώ. Η παρουσίασή σας ήταν περισσότερο μια ωραία ιστορία δημοσίων σχέσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ε, υποστηριζώ απόλυτα. Αναφερθήκατε στο 2017, το οποίο συζητάμε εδώ. Με μεγάλη μας χαρά σας ακούσαμε και χαιρόμαστε που μαθαίνουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας ε, είναι ουσιαστικά ε, παρέχει μια, μια υπηρεσία. Χαίρομαι γι' αυτό υπογραμμίσατε σε επιδόσεις και είπατε ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα για το επόμενο μακροχρόνιο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ λέγει εδώ το 2009. Τότε δεν συζητούσε πολύ ο κόσμος την απόδοση, όχι εδώ τουλάχιστον, ούτε καν στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά έχουν αλλάξει πολλά έκτοτε. Χαίρομαι που υπογραμμίζετε την απόδοση, αλλά αν δω την ανακοίνωση στην οποία βασίζεται η σημερινή συζήτηση ε, με τους ετήσιους λογαριασμούς ε, στο προήμιο του Επιτρόπου Έτιγκερ ε, και μόνο η τελευταία οι κάθε δύο προτάσεις αναφέρουν σε απόδοση και φυσικά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι σημαντική αλλά για μένα η απόδοση έπρεπε να είναι το κεντρικό σημείο όχι μόνο όταν κάνουμε δημόσιες σχέσεις αλλά και όταν κάνουμε πραγματική δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλετε να πούμε δημοσίως τι ωραία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πείτε πόσο αποτελεσματική είναι, την αποτελεσματικότητα της, την απόδοσή της. Έτσι μπορούμε να δείξουμε στους λαούς της Ευρώπης ε, ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης πραγματικά να ξέρουν ότι δεν ε, ε, έχουμε απλά ποσά να κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι επενδύουμε πραγματικά στου τομεί υψηλότερη προστιθέμενη αξία και όπου πραγματικά βλέπουμε αποτελέσματα και καλέ επιδόσει. Όπω είπατε, οι επιδόσει, η απόδοση είναι ένα βασικό στοιχείο στην πρόταση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Εγώ διάβασα πολύ προσεκτικά την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου τη 7η Νοεμβρίου για την Γεωργία και για την κοινή γεωργική πολιτική. Αν η κοινή γεωργική πολιτική έχει κάποια χαρακτηριστικά, ε, η απόδοση δεν είναι από αυτά, δεν βασίζεται σε αυτά. Αυτό λέει το μήνυμα του Ελεκτικού συνεδρίου. Έχετε προειδοποιηθεί ήδη πριν από την πρόταση για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Πριν από ένα χρόνο το ελεγκτικό συνέδριο είχε εκδώσει μια έκθεση για το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής και εκεί σας προειδοποιούσαν ε, για την απόδοση, ότι αν λάβετε την απόδοση ως βάση πρέπει να αλλάξετε ριζικά την πολιτική. Και α είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, τίποτα δεν άλλαξε ριζικά. Και το βασικό μήνυμα του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι οι άμεσες ενισχύσεις εξορισμού δεν βασίζονται στις επιδόσεις. Θα μπορούσατε να το σκεφτείτε λίγο αυτό. Για να μην μιλάμε μόνο για το έτος 2017. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, κάτι που ήθελα να πω Όλοι αυτοί οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και ειδικότερα σε πρώην, ε, πρώην γενικοί διευθυντέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, αυτό συμβαίνει. Μετά αναλαμβάνουν κάποια ιδιαίτερα καθήκοντα, γίνονται ειδικοί σύμβουλοι. Εδώ στο χαρτί μου βλέπω ότι το 2017 υπήρχαν 118 ειδικοί σύμβουλοι. Από όσο γνωρίζω, όλοι αυτοί οι 118 δεν είχαν τόσο σημαντικά καθήκοντα που να εστιάζονται υπερβολικά στην προστιθέμενη αξία. Ξέρω ότι πολλοί από αυτού περνάνε πολύ χρόνο στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο τη Φλωρεντία. Εμένα δεν με πειράζει που είναι συχνά στη Φλωρεντία, αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε τι τεράστιε γνώσει και την εμπρογνωμοσύνη του καλύτερα. Πολύ καλύτερα, μάλιστα, για να δημιουργήσουμε πολύ υψηλότερη προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η ερώτησή μου για το 2017 και για την ε, πολιτική προσωπικού κύρια. Πρόεδρε, δυστυχώς έχω να ψηφίσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά ε, το προσωπικό μου θα λάβει σημειώσεις ε, για τις απαντήσεις του κυρίου Γενικού Γραμματέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Σελμάιερ. Δεν έχουμε συναντηθεί και Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να κάνουμε μια προσωπική συζήτηση μεταξύ μας. Έχω διάφορες ερωτήσεις. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και απόδοσης. Είναι η δική σας αξιολόγηση για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των πραγμάτων. στο πλαίσιο του συντονισμού του, του γραφείου σας, ε, του Γενικού Γραμματέα. Διαβάζοντας την έκθεση βλέπω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Λέει ότι τα σημαντικότερα πράγματα που έχει κάνει η Κομισιόν ε, λέει ποια είναι, ποιοι είναι οι συντελεστέ σφάλματος, ε, οι οποίοι φαίνεται να είναι πολύ καλοί. Αυτή είναι η δική σας αξιολόγηση, η δική σας αποτίμηση, ή έχει εμπλακεί και το ελεκτικό συνέδριο. Το έχει κοιτάξει, το έχει ελέγξει. Το ελεκτικό συνέδριο προλαβαίνει. Έχει χρόνο να αφιερώσει για να ρίξει μια ματιά σε αυτή την έκθεση, να τη διαβάσει ε, εξονυχιστικά, να εντοπίσει πράγματα που χρήζουν περισσότερη προσοχή, να δει πράγματα που ίσω δεν είναι σωστά, που πρέπει να διορθωθούν. Εγώ το διάβασα με του συναδέλφου μου και παρατηρώ ότι αν δει τη σύνοψη της οικονομικής διαχείρισης στην έκθεση αυτή, λέει ότι εσείς ως Επιτροπή αναφέρει το 1,7% και αυτό είναι μια χαρά, αλλά στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου του 2017 αυτό είναι το ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές από όσο φαίνεται. Τι λέτε λοιπόν ότι αυτό το 1,7% με αυτό το 1,7% εξακολουθούμε να είμαστε κάτω από το 2% του περιθωρίου ουσιοδός σφάλματος οπότε πάμε καλά. Αλλά αν δω την έκθεση του ε, ελεκτικού συνεδρίου του 2017, εκεί παρατηρώ ότι το ελεκτικό συνέδριο αναφέρει πολλές αδυναμίες, πολλά σφάλματα, ειδικότερα όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα. Και εκεί αναβαίνουμε πάνω από το 2%. Λέει για παράδειγμα ότι η Κομισιόν δεν έχει ένα άλλα 13 διαφορετικά περιθώρια ασφάλματο και ότι τα περιθώρια ασφάλματο δεν είναι οριστικά γιατί όπως φαίνεται έχουν υπολογιστεί σε σχέση με πιστώσει. με δεσμευμένες πληρωμέ. Ε, και όπως φαίνεται αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά το οικονομικό μέσο και μπορεί το αποτέλεσμα το τελικό να είναι διαφορετικό ε, ήθελα να μου πείτε λοιπόν τη δική σας άποψη. Πώς γίνεται η δική σας έκθεση να είναι τόσο διαφορετική από εκείνη του ελεγκτικού συνεδρίου. Άλλες ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω είχαν ως εξής. οι προσαρμοσμένοι κανονισμοί για τα δημοσιονομικά, οι συζητήσεις για την ΚΑΠΑ, ο κανονισμός για τις κοινέ διατάξεις, σχετικές διαπραγματεύσεις. Τι γίνονται με τους ελέγχους που κάνει η Κομισιόν για τις πληρωμές, ε, ε, έχουν μειωθεί, ε, τους έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη. Φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες, έτσι υπόθηκε στο πλαίσιο αυτό. Έχω ερωτήσει λοιπόν γι' αυτό. Όπως έμαθα, είναι και μεγαλύτερε οι προσδοκίε των κρατών μελών. Και αυτό έχει ληφθεί υπόψη στις εθνικές νομοθεσίες, οικονομικές πτυχές. Ποια είναι η ιδεολογία. είμαι περίεργο. Διότι αν είναι να διαβιβάσετε έλεγχο από το κεντρικό στο εθνικό επίπεδο, δηλαδή να εκχωρήσετε αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Πώς αναμένεται σε κράτη-μέλη με ελλειπές κράτος δικαίου και ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Σε τέτοια κράτη λοιπόν πώς μπορούμε να αναμένουμε ότι θα αναλάβουν ελέγχους ε, ε, και θα τους πραγματοποιήσουν αρκετά ικανοποιητικά ώστε να παραμείνει ε, το ποσοστό σφάλματος κάτω από το όριο. Αυτή είναι η δεύτερη συνερωτήση που θέλω να κάνω. Και μετά τι γίνεται με την κατάσταση της τσεχικής δημοκρατίας. Το, αυτό το πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα. Πολλοί επίτροποι έχουν ερωτηθεί γι' αυτό. Έγινε και μια επίσκεψη στη τσεχική δημοκρατία. Ε, ε, συνέβησαν διάφορα περίεργα εκεί. Υπήρξε μια καταγγελία της διεθνούς διαφάνειας ε, στην τσεχική δημοκρατία. Υπήρξε μια ανταλλαγή ε, επιστολών, υπήρξαν κάποια θέματα με το κόμμα των πειρατών, υπήρξε η κατάσταση που αφορά τον Πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας, ο οποίος ε, είναι ύποπτος ε, διαφθοράς και τα λοιπά και ότι υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της θέσης του και τη σχέση του με μια επιχείρηση που λαμβάνει ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις εκατομμυρίων. Στην Επιτροπή λοιπόν Ελέγχου του Προπολογισμού έχουμε πολλά ερωτήματα για τα θέματα αυτά. Έχουμε συζητήσει με τον Επιτροπό Ετίνγκερ το Σεπτέμβριο και μα απάντησε ότι η Κομισιόν το παίρνει αυτά πολύ στα σοβαρά και ότι θα πραγματοποιηθούν κοινέ έρευνε ε, και με όλες τις ε, εμπλεκόμενες γενικές διευθύνσεις. Πριν από τρεις εβδομάδες στο Στρασβούργο, αυτό επικυρώθηκε και από τον Επίτροπο Χόγκαν ότι γινόταν μια κοινή έρευνα από την Άγκρη, Ρίτζο ε, και Μπάτσε. Και οι τρει ε, ενεπλάξαν σε αυτή την κοινή ε, έρευνα και χθε εδώ ήταν η κυρία Κρέτσου και στι γραπτέ τη απαντήσεις ερωτήσεις μα για το ζήτημα αυτό ειδικότερα είπε ότι δεν υπάρχει επίσημη κοινή έρευνα. Ναι, ερευνάμε. Βάσει μιας καταγγελίας που έχει υποβληθεί. Αυτή η απάντηση είναι ίδια με τη δική σας. Ναι, σε κάποιο βαθμό. Ε. Στη γραπτή σας απάντηση δεν λέτε ότι υπάρχει κοινή έρευνα, απλά λέτε και εσεί, θα μας ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνο για την κατάσταση, αλλά δεν αναφέρετε τίποτα για κοινή έρευνα. Σήμερα το απόγευμα είχαμε μια συνάντηση με τους γενικούς Διευθυντέ και του αρμόδιου στην Apple, στην Άγκρη, στη Ρίτζο και στην τέταρτη γενική διευθυνσή που εμπλέκεται και όπως φαίνεται οι γενικές διευθύνσεις πραγματοποιούν έρευνα και συντονισμένα μάλιστα. Πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι γίνεται έρευνα, κοινή έρευνα. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και είναι συντονισμένη κοινή έρευνα μεταξύ τεσσάρων ε, γενικών διευθύνσεων και μετά Ξέρετε, πολύ συχνά, η Κομισιό, πολύ σύντομα η Κομισιόν θα χρειαστεί να μας παρουσιάσει και τα αποτελέσματα αυτής της κοινή έρευνας εδώ στο Κοινοβούλιο. Εδώ μιλάμε για σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ Πρωθυπουργού και μιας εταιρείας την οποία ή ελέγχει ή την ήλεγχε κτλ. τα θέματα δεν είναι μόνο θέματα δηλαδή του κανονισμού για τα δημοσιονομικά, του οικονομικού κανονισμού, αλλά σήμερα μας είπαν ότι ο προηγούμενος τέτοιος κανονισμός, ε, ο προηγούμενος financial regulation και άλλοι κανονισμοί και άλλα νομικά μέσα περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες ε, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, καταστάσεις. Θέλω να ακούσω λοιπόν και τη δική σας άποψη κύριε Γενική Γραμματέα γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό πράγματι. ο κόσμος είναι πολύ ευαισθητοποιημένος, ειδικά στην Τσεχική Δημοκρατία έχουν γίνει κοινοτοποίησεις, θα ψηφιστεί, θα υπάρξει μια ψηφοφορία το Σάββατο στο Τσεχικό Κοινοβούλιο. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε θα μας ήταν ωφέλιμο. Ευχαριστώ. Άλλοι τρει ομιλητέ, ο κύριος De Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω πως τουλάχιστον εγώ προσωπικά θα ήθελα να ευχηθώ. Καλώς ορίσατε στον κύριο Σελμάγερ έχουμε ακούσει πολύ συχνά να μιλάνε για σας και για το διορισμό σας. Να πω πως από τη συζήτηση που γίνεται εδώ πρέπει να σας πω πως ήταν η διαδικασία ε, διορισμού η οποία συζητήθηκε και όχι η ποιότητα της υποψηφιότητας σας και εύχομαι να συνεργαστούμε σωστά και αποτελεσματικά στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να συνταχθώ με τα όσα είπε ο Γενικός ε, Γραμματέας. Χτες τα είπαμε πολύ λεπτομερώς στην έκθεση για τους νέους ε, κανόνες ε, για το διορισμό των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είδαμε πως υπάρχουν πολλά στοιχεία προόδου όσον αφορά την ακαιρεότητα. Θα είμαι, εν ή σύντομος, κυρία Πρόεδρε γιατί πρέπει να έχουμε και χρόνο για να ακούσουμε τις απαντήσεις. Η θέση οριζόντια για την εκείνη τη διαδικασία προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πείτε μου τι θα γίνει. Έχουμε το ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μήπως θα είναι ο διαμεσολαβητής ο οποίος θα μπορούσε να είναι το σημείο προς το οποίο θα φεύγει η κοινοποίηση. Και αυτό σε περίπτωση που έχουμε, για παράδειγμα, κάποια καταγγελία για τα που να θέτει σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Και τι θα μπορεί να κάνει ο καθένας εκτός του δικού του περιορισμένου επαγγελματικού πλαισίου, έτσι ώστε να προχωρήσουμε Και για τους καταγγέλλοντες ε, θα ήθελα να μου πείτε Ε, τι γίνεται με την Woolly Post, η οποία δούλευε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απολύθηκε το Σεπτέμβριο γιατί θεωρήθηκε πως έχει ε, προβεί σε καταγγελία, δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες της συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πριν απολυθεί κάποιο αυτό θα πρέπει να εξετάζεται, γιατί ξέρετε πω τουλάχιστον στην Βουλή ε, της, ε, των κάτω χωρών και στον τύπο στη χώρα μου ε, συζητήθηκε πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή κρύβεται κάπου στην Ολλανδία. Και έχουμε ένα αίτημα και έχουμε ένα αίτημα από πλευράς Ευρωπαϊκή, ε, ε, Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που ζητά να επιστραφούν 190.000 ευρώ. Όχι, λοιπόν, ότι ξέρω όλο το θέμα, αλλά με ενδιαφέρει και η ανθρώπινη διάσταση. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες, δεν ζητώ κάτι άλλο, αλλά απευθύνομαι προς τη Γενική Διεύθυνση ε, που την ε, κυνηγά, αλλά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος καταγγέλει θα πρέπει να προστατεύεται με κάποιο τρόπο και θα πρέπει να το χειριζόμαστε διαφορετικά, ε, ειδικά όταν είναι υπάλληλοι μας. Το έχω, μιλή, το έχω συζητήσει και με τον ε, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ατύπους. Θέλω να το κάνω τώρα και δημόσια, να βρούμε μια καλή λύση για το άτομο αυτό. Δεν πρόκειται να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα μας βοηθήσει πολύ Ε, για όλα αυτά τα θέματα που άπτονται του νέου κανονισμού. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με, τις, ε, με τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω ε, τον Γενικό Γραμματέα αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο που βρίσκονται εδώ σήμερα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία απαλλαγή για τον προπολογισμό του 2017 και εδώ έχουμε πολιτική ευθύνη, έχουμε δημοκρατική, δημοκρατικό έλεγχο και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έρχονται ε, και η Επιτροπή. Είχαμε χθε την Επίτροπο Περιφερειακής ανάπτυξη, σήμερα το πρωί τον Επίτροπο κύριο Μίντα. Καλό είναι που έχουμε και το Γενικό Γραμματέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής εδώ μαζί μα για να έχουμε μια αμοιβαία κατανόηση για τα θέματα που μα αφορούν. Η συνεργασία μεταξύ θεσμών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να γίνονται με αρμονικό τρόπο έτσι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα να προχωράει. Εγώ δεν πρόκειται να αναφερθώ στο διορισμό του Γραμματέα εγκρίθηκε το ψήφισμα από την Ολομέλεια και θα συζητήσουμε τη συζήτηση αυτή και στα πλαίσια της Επιτροπής ε, Εσωτερικού Κανονισμού στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να πω προς το Γενικό Γραμματέα πως έχουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι ιδέες έχει για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες ε, μέσα στο όργανο αυτό. Επίσης, ένα σημείο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η επικοινωνία. Πώς μπορούμε δηλαδή να βελτιώσουμε την επικοινωνία και προς το όργανο αυτό στη πλαίσια της προσπάθειας διαφάνειας και βελτίωσης της φήμης που έχουν τα δικά μας όργανα ε, στα μάτια του πολίτη. Δεν είμαστε απάτριδες ε, γραφειοκράτες όλοι, απρόσωποι. Είμαστε άνθρωποι και επειδή διάβαζα το ερωτηματολόγιο σε βάθο, θα ήθελα να δω πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τη φήμη μα, το πώ μα βλέπουν. Είναι ένα κομβικό όργανο στο ευρωπαϊκό οικοδόμα. Και δύο τελευταίε ερωτήσει όταν μπήκα στην ε, συνάντηση, ο Γενικό Γραμματέα μιλούσε για τη σημαντική συμφωνία που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα όσα έκανε στα πλαίσια τη εμπορική πολιτική και όταν, ε, όταν ε, κατέρευσε η, η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε Καναδά, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Περνάμε λοιπόν ε, αυτή τη στιγμή και μια πολύ κρίσιμη στιγμή γιατί μιλάμε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Έχουμε μια ε, συνάντηση αυτή την εβδομάδα και μια υπουργική η οποία αναβλήθηκε. Τι γίνεται λοιπόν. Έχετε λάβει όλα τα μέτρα για να συντονιστείτε με τις υπόλοιπες γενικές διευθύνσεις. Ε, για το τι θα γίνει. Γιατί είναι μια τεράστια αγορά 450 ε, εκατομμυρίων ανθρώπων και νομίζω ότι θα δείξει και ποιε είναι οι προθέσει μα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πούτε αν οι γενικέ διευθύνσει σα έχουν συντονιστεί. Τέλο, χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Είμαι εισηγητή στην ΑΦΕΤ για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πολύ σημαντικό, 14 δις ευρώ και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η θέση σας για την φύση τη μοναδική φύση αυτών των ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων. Γίνεται η συζήτηση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέσεις πολύ σαφείς υπέρ ενός τέτοιου μοναδικού εργαλείου, αλλά κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν πιστεί για το ότι χρειάζεται. Αυτό το οποίο εγώ πιστεύω είναι τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου στην παρακολούθηση των χρηματοδοτικών εργαλείων να διατηρηθούν και θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύει ο Γενικός Γραμματέας για αυτό το θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση σε πολλές επιτροπές και το οποίο είναι τόσο σημαντικό. Πυρίνσκι, τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι κι εγώ όσο το δυνατόν περισσότερο σύντομος. Κύριε Γενική Γραμματέα, θέλω να πω ότι Πιστεύω ότι η ακαιρεότητα είναι μια διαδικασία που βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας απαλλαγής και πιστεύω ότι εδώ και τώρα πρέπει να μας δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά σημεία που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18 Απριλίου και να αναφέρω τρία σημεία από αυτά. Μήπως προσπαθήσετε να τα απαντήσετε. Το πρώτο είναι γιατί χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφορετικές διαδικασίες ε, για τον διορισμό του Γενικού ε, ε, Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στην ίδια συνεδρίαση. Είπατε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες. Γιατί ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικοί κανόνες από ό,τι φαίνεται. Τώρα, λίγο έξω από το, δικό σας, το θέμα του δικού σας διορισμού, ζητήθηκε να επανεξεταστεί με βάση το άρθρο 29 ο διορισμός των ανατάτων στελεχών με το στόχο να διασφαλίσουμε ότι επιλέγονται οι καλύτεροι υποψήφοι μέσα σε ένα πλαίσιο της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών δίνοντας το υπόδειγμα για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και στην παράγραφο 30 αναγνωρίζουμε ότι ε, το άρθρο 17 δίνει ιδιαίτερες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα που πρέπει να έχει και εμπειρία διοίκησης και την εμπιστοσύνη του Προέδρου και πρέπει να είναι σαφές ότι θα, θα επικαιροποιούνται οι κανόνες για να είναι εγγυημένη η ουδετερότητα του Γενικού Γραμματέα και αναμένεται ότι θα ενημερώνεται μέχρι το Σεπτέμβριο του 2018 για τα αποτελέσματα αυτά. Θα ενημερώνεται δηλαδή το Κοινοβούλιο. Αν μπορείτε παρακαλώ θα σας ήμουν ευγνώμων να μας απαντήσετε. Πολλές ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών για τις ε, σοφές ερωτήσεις ε, που έχετε θέσει και θα ξεκινήσω από το τέλος που είναι οι πιο δύσκολες ερωτήσεις για μένα και εγώ άνθρωπος είμαι θα έλεγα μην αμφισβητείτε την ακεραιότητά μου, γιατί αν αμφισβητείτε την ακεραιότητά μου δεν με γνωρίζετε. Και αυτό το λέω γιατί ποτέ δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία να πω τίποτε από αυτού. Μην αμφισβητείτε την ουδετερότητά μου. Αν, αν έχετε ε, κάτι εναντίον μου να μου το πείτε. Δεν είμαι κομματικός. Αν ακούτε φήμες, οι φήμες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια καλύτερα να μιλάτε με τους ανθρώπους και όχι γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι καλύτερα να συζητάτε με τον ενδιαφερόμενο παρά ε, να μιλάτε για τον ενδιαφερόμενο. Μετά από 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ολόκληρη τη ζωή μου που αφιέρωσα στην οικοδόμηση της Ευρώπης, δεν πρέπει να αμφισβητείτε την ουδετερότητά μου και την ακαιρεότητά μου όταν κρίνετε κάποιον πρέπει να ακούτε τον ίδιο αυτό τον άνθρωπο. Η απόφαση λήφθη από το Σώμα των Επιτρόπων και χαίρομαι διότι ως άτομο εγώ χαίρομαι γιατί επελέγει από το Σώμα των Επιτρόπων βάσει μιας διαδικασίας. Θα μπορούσε το Σώμα των Επιτρόπων να με διορίσει απλώς, αλλά πέρασα μέσα από μια διαδικασία όπου απέδειξα τι μπορώ να κάνω. Πάτε στην ερώτησή σας τι εμπειρία διοίκηση έχω είτε είμαι ανίκανος και δεν μπορώ να διοικήσω, είτε διοικώ τα πάντα. Δεν μπορεί να, λέτε, να λένε στις Βρυξέλλες και ότι είμαι ανίκανος και ότι διοικώ τα πάντα. Έχω αποδείξει σε όλες τις διαδικασίες, στα 40 χρόνια επαγγελματικής μου καριέρας, ε, ποια είναι η εμπειρία μου. Αν έχετε όμως τη στοιχεία ότι δεν μπορώ να διοικήσω, ελάτε στην Επιτροπή και να μας το πείτε. Αλλά να μην μιλάμε για φήμες. Η Επιτροπή δεν ακολούθησε διοικητικέ διαδικασίε, ακολούθησε νομικέ διαδικασίε βάσει του κανονισμού προσωπικού. Δεν είναι εσωτερικοί οι κανόνε τη Επιτροπή, είναι κανόνε που έχουν θεσπίσει οι νομοθέτε. Και η ίδια διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί πολλέ φορέ για πολλά άλλα άτομα στην Επιτροπή, αλλά φαίνεται πρόβλημα να έχετε μόνο με μένα. Παραδεχτείτε το ότι έχετε πρόβλημα μαζί μου και όχι με τι διαδικασίε. Αν έχετε πρόβλημα μαζί μου, πείτε μου ποιο πρόβλημα έχετε μαζί μου, αλλά κανεί δεν τολμά να μου το πει. Δεν είμαι τέρα, ανθρώπινο όνειμα κι εγώ και ευρωπαϊστή. Οπότε οφείλω κι εγώ να ναι, έχω το δικαίωμα να απολογηθώ. Η κυρία Γκρέσλε μίλησε ε, για το θέμα των απαντήσεων στις κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις. Κάποιος, ε, ε, εγώ ίδιος είμαι κάποιος που παίρνει ιδιαίτερα στα σοβαρά αυτά τα θέματα. Διαβάζω όλες τις ερωτήσεις, τις γραπτές κοινοβουλευτικέ ερωτήσεις και προσπαθώ να δίνουμε την καλύτερη δυνατή απάντηση. Βέβαια είναι τεράστιο ο αριθμός και γι' αυτό ζητώ συγγνώμη αν δεν είναι πάντοτε τέλειες οι απαντήσει, αλλά προσπαθούμε να βελτιώνουμε τις απαντήσεις μας. Δεν απαντώνται από το Γενικό Γραμματέα βέβαια οι ερωτήσεις. Οι Επίτροποι και τα Γραφεία των Επιτρόπων εξετάζουν τις ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής διαδικασίας από το Σώμα των Επιτρόπων. Αλλά μπορεί καμιά φορά να, να μην είναι μια ξεκάθαρη απάντηση όπως θα έδινε ένας Επίτροπος μια ξεκάθαρη απάντηση, απάντηση επιτόπου. Ε, κάθε γραπτή απάντηση δεν πηγαίνει μόνο σε έναν Επίτροπο, περνάει από όλο το Σώμα των Επιτρόπων. Πάντως αποδίδω μεγάλη σημασία, τις θεωρώ πολύ σημαντικές και μπορείτε να βασίζεστε σε μένα σχετικά αυτό. Για το θέμα των στατιστικών δεδομένων. Είπατε ότι υπάρχουν αμφιβολίες για την συνέπεια των στατιστικών ε, στοιχείων. Εν μέρη συμφωνώ και πριν από λίγες εβδομάδες ε, στείλαμε μια επιστολή προς όλες τις υπηρεσίες της Eurostat για να βελτιώσουν την ε, ποιότητα γιατί χρειαζόμαστε αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα τα οποία αποτελούν βάση για τις πολιτικές μας. Ρωτήσατε επίσης κυρία Πρόεδρε, για ε, την Επιτροπή ε, Ελέγχου, την Audit Progress Committee. Αυτή η Επιτροπή ε, αποτελεί από μόνη της μια τεράστια βελτίωση για την Επιτροπή μας, διότι σε κάθε συνεδρίασή τους υπάρχει κάποιος επίτροπος. Και ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμαντς παίρνει ιδιαίτερα σοβαρά την όλη αυτή η διαδικασία. Στο παρελθόν δεν παρευρίσκονταν οι επίτροποι. Εδώ κάθε φορά παρευρίσκονται 4-5 επίτροποι και γενικοί διευθυντέ. Δηλαδή η διαδικασία είναι κατά πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Και το τι θα κάνουμε με τη δέσμη εταιρική διακυβέρνηση, αν εγκριθεί αύριο από το Σώμα των Επιτρόπων. Και βέβαια θα σας δοθούν τα έγγραφα αυτά για να τα μελετήσετε. και η όλη διαδικασία θα ενισχυθεί για την συνεργασία με το Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης. Εμείς δεχθήκαμε όλες τις συστάσεις ε, της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητη, και ελπίζω θα σας ικανοποιήσουν και εσάς οι απαντήσεις μας. Για τις περικοπές προσωπικού ε, κατά 5%. Εγώ ήρθα στην Επιτροπή από τον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η καλύτερη δημόσια υπηρεσία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όλοι οι υπάλληλοι δουλεύουν σκληρά με τον νέο κανονισμό προσωπικού μπορεί να μην έχουν καταλάβει ε, οι πολίτες εν γέννη πόσες ώρες δουλεύουν ε, οι υπάλληλοι της Επιτροπής. Αν δείτε την, ε, τις συμφωνίες που συνάπτουμε, τα, τις ώρες που έχουν μπει για τη Συμφωνία Μερκοσούρη για τον Brexit, είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο ρυθμός των ωρών. Όντω υπήρξε η δημοσιονομική κρίση και γι' αυτό κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έπρεπε να εξετάσουμε όλε τι πτυχέ των εθνικών πολιτικών. Το θέμα της μετανάστευσης. Ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εν μέρη υπεύθυνη, όχι νομικά υπεύθυνη, αλλά πολιτικά υπεύθυνη να βοηθήσει στα ελληνικά νησιά, να βοηθήσει για τη διοίκηση και διαχείριση της μετανάστευσης στα κράτη-μέλη. συνεχίσαμε με περικοπές προσωπικού να αναβαθμίζουμε τις εργασίες μας με υψηλότερη ε, ποιότητα ε, προσωπικού και με υψηλότερες υπηρεσίες τις οποίες ε, αποδίδουμε. Έγινε και κάποια ερώτηση για τους συμβούλους. Δεν νομίζω ότι παρακάμψαμε τον κανονισμό προσωπικού, γιατί προβλέπεται στον κανονισμό προσωπικού αυτό. Ο κανονισμό προσωπικού περιέχει πολλά διαφορετικά μονοπάτια καριέρα. Ένα μονοπάτι πηγαίνει στην ε, διοίκηση. Κάποιοι είναι πολύ καλοί ω σύμβουλοι, έχουν την ικανότητα να κάνουν κάτι άλλο. Είναι εμπειρογνώμονε και μπορούν να πάρουν κάποιες, ε, κάποια προαγωγή ε, ω εμπειρογνώμονε. Είναι πολύ λογική η οργάνωση τη Επιτροπή και ο κανονισμό του προσωπικού ανοίγει αυτά τα μονοπάτια καριέρα που τα χρειαζόμαστε γιατί χρειαζόμαστε και τα δύο και συμβούλου και ε, ε, στελέχη που μπορούν να διοικήσουν. Αναφέρεται και το EPSC που είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο ε, είχαμε στην προηγούμενη Επιτροπή. Στην παρούσα Επιτροπή, το EPSC είναι άτομα που συμβουλεύουν τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους στο συντονισμό και διαχείριση προγραμμάτων και μερικές φορές κοιτάζουν και πιο μακροπρόθεσμα πέρα από την καθημερινή δουλειά που γίνεται στην Επιτροπή εξετάζουν την Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το οποίο δημοσιεύθηκε παραδείγματος χάρη πέρυσι ε, το Μάρτιο, το 2018 το Μάρτιο δεν ε, ε, προγράφουν το μέλλον της Ευρώπης, αλλά εξετάζουν διαφορετικούς τομείς στους οποίους, προς μπορεί να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύουν και με τις ομάδες έργου για την παγκοσμιοποίηση, για τον κοινωνικό τομέα, σε πάρα πολλούς τομείς. Και μην νομίζετε ότι είναι παιδιά και ανήψια ε, υπαλλήλων της Επιτροπής. Ε, ισχύει αξιοκρατία και έχουν προσληφθεί μόνο με βάση τα προσόντα τους και ο επόμενο πρόεδρο, το επόμενο κολέγιο μπορεί να αποφασίσει να προσλάβει άλλου ανθρώπου. Οι συμβάσει του τελειώνουν στο τέλο τη θητεία αυτή τη Επιτροπή, όπω συνέβη και στην προηγούμενη Επιτροπή, όπου κάποιοι είπαν Μα αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν απολυθεί από την Νέα Επιτροπή. Ε, δεν είναι αλήθεια, δεν απολύθηκαν από την Νέα Επιτροπή, απλά έλξαν οι συμβάσει του. Ο κ. Γκερμπράντι δεν είναι εδώ, ε, αλλά οι συμβουλοί του θα του το πούν ε, όσα θα πω τώρα. Όταν μιλάμε θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο θέμα δημοσίων σχέσεων. Πρέπει να το κάνουμε βάσει στοιχείων. Όταν υπάρχουν στοιχεία, πρέπει να αναφέρονται. Καμία δημόσια σχέση αβάσιμη δεν είναι βιώσιμη. Πάντα πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία. Εγώ δεν βλέπω μεγάλη διαφορά μεταξύ της ετήσιας εκθεσής μας ε, απόδοσης της διαχείρισης και των συμπερασμάτων του ελεκτικού συνεδρίου σύμφωνα με τα στοιχεία. Ναι, δείχνουμε μια θετική εικόνα, όχι υπερβολικά θετική, είμαστε ρεαλιστέ. Αλλά ναι, καταφέραμε κάποια πράγματα το 2017 και το ελεκτικό συνέδριο φυσικά ω ελεγκτέ έχουν ένα άλλο στυλ. Λένε σε γενικέ γραμμέ, ναι, σε μεγάλο βαθμό η Επιτροπή χρησιμοποίησε με αποδεκτό τρόπο τα χρήματα των, χρηματο... των φορολογουμένων. Γι' αυτό έδωσε ε, καλή ε, γνωμοδότηση για δεύτερη φορά συνεχή δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίφαση. Ίσα ίσα που είμαστε σύμφωνοι και αυτό είναι καλό. Γιατί αλλιώ θα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά περισσότερα ω αντίδραση στη συστάση του ελεκτικού συνεδρίου για του ε, συμβούλου, 118 ε, ειδικού συμβούλου που αναφέρατε. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οι ειδικοί σύμβουλοι ε, συμβουλεύουν του ίδιου του επιτρόπου. Οι περισσότεροι από αυτού δεν πληρώνονται. Ε, λαμβάνουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Υπάρχουν κάποια άλλοι σε ανώτερες θέσεις στην Κομισιόν που γίνονται ε, σύμβουλοι υψηλή, υψηλόβαθμοι έχουν ε, υπηρετήσει ω γενικοί διευθυντές αλλά στα τελευταία του χρόνια στην Κομισιόν παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη χωρίς τα διοικητικά. Έχουμε το Γενικό Διευθυντή της DigiHome που υπήρξε Γενικός Διευθυντής για πολλά χρόνια και βοηθά το Γενικό Γραμματέα ε, με συμβουλευτική υποστήριξη για το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο, για τη μετανάστευση στο μέλλον, για τα θέματα μεταφορών και για τα ζητήματα ετοιμότητας για τον Brexit. Και όλα αυτά είναι πολύ καλά. Δεν πρέπει να χάνουμε τους ανθρώπους που έχουν συγκεντρώσει τόσο τεράστια εμπειρία την τελευταία χρόνια απλά τι θητείε του, του λέμε να μην κάνουν διοικητικά καθήκοντα και να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη. Και αυτό δεν του ε, ε, δυσαρεστεί καθόλου. Είναι μια κατάσταση υποφελής προς όλους. Δεν περνάνε χρόνο στη Φλωρεντία. Αν κάποιο έχει πάει στη Φλωρεντία είναι γιατί έχουμε εκεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο κύρος παγκοσμίω και μερικές φορές μας δίνει πολύ καλά αποτελέσματα και στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή που συνεργάζονται στενά. Κυρία Στάς, αναφέρατε πολλές σημαντικές ερωτήσεις. Να τις δούμε με τη σειρά αισιόδοξη άποψη, μιλήσατε για την ετήσια διαχείριση. Ναι, έχουμε ετήσια, ε, αισιόδοξη άποψη. Είδαμε ότι μετά από πολλά χρόνια κρίση και δυσκολιών καταφέραμε μαζί σα και με το Συμβούλιο να τα καταφέρουμε αρκετά καλά το 2017. Και ε, με τα εξωτερικά αποτελέσματα αυτό είναι προφανέ. Ε, το βλέπουμε και στην εκθέση του Ελεκτικού Συμβουλίου, παρότι σε ορισμένα σημεία είναι πιο επικριτική. Κάποιε διαφορέ στα νούμερα, όχι επί τη συνολική αξιολόγηση, Κάποιε διαφορέ ε, υπάρχουν γιατί άλλε φορέ κοιτάμε τα νούμερα ε, σε αιτήσιο πλαίσιο ή σε πολιτέ πλαίσιο και εκεί φυσικά υπάρχουν διαφορέ στα νούμερα. Έχει να κάνει με την πολύπλοκη φύση του πολιτού δημοσιονομικού πλαίσιου. Έχουμε προσπαθήσει τι προτάσει μα, όπω τι προτείναμε τον Μάιο και τον Ιούνιο, Έχουμε προσπαθήσει μέσα αυτών των προτάσεων να υπέρθουν κάποιε απλουστεύσει, να εστιαστούμε περισσότερο σε επιδόσει, όπω είπε και ο κ. Γκερμπράντι. Διότι το βασικό μας θέμα εδώ είναι η προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωση και οι επιδόσεις και ελπίζω οι συνομοθέτες να μας υποστηρίξουν. Σα ευχαριστώ για την ενδιάμεση σα έκθεση γι' αυτό γιατί πολλά από τα λόγια που χρησιμοποιήσατε εκεί πέρα μας βοήθησαν. Επίσης ρωτήσατε για την κοινή γεωργική πολιτική και τη μεταρρύθμιση τη. Υπάρχει τίποτα άριστο. Έχουμε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και εγώ δεν θα διαφωνήσω. Είναι ευκολότερο να την επικρίνει κανεί παρά να τη βελτιώσει. Φυσικά η κοινή γεωργική πολιτική είναι η παλιότερη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τι οποίε ε, υποστηρίζεται και για την οποία είναι περήφανα πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μα ευχαριστούν για αυτή. Η Κομισιόν με την πίεση του Επιτρόπου Χόγκαν έχει προσπαθήσει να εξυγχρονίσει την πολιτική αυτή χωρί να την να κάνει επαναστατικέ αλλαγέ. Ένα στοιχείο είναι να αναθέσουμε περισσότερε ευθύνε στα κράτη-μέλη να εκχωρήσουμε περισσότερε ευθύνε, όπω έχει ζητηθεί από πολλού από εσά και σε αυτή την επιτροπή και σε άλλε. Όχι γιατί θέλουμε να ξεφορτωθούμε τον έλεγχο. Σίγουρα όχι. Απλά πιστεύουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει είναι προτιμότερο η διαχείριση κάποιων πραγμάτων να γίνεται επί τόπου. Η κοινή γεωργική πολιτική ήδη βρίσκεται υπό επιμερισμένη διαχείριση. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό σημαίνει ότι εμεί πρέπει να ε, τα δώσουμε όλα στα κράτη-μέλη. Είπατε ότι υπάρχουν κάποια θέματα με το κράτο δικαίου. Με το κράτο δικαίου συμφωνώ μαζί σας και εγώ υπερασπίζομαι το κράτος δικαίου όχι μόνο γιατί είμαι νομικός αλλά γιατί πιστεύω ότι το κράτος δικαίου είναι ε, αυτό που κραταδεμένη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είμαστε τόσο αφοσιωμένοι σε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν είπα ότι θα πραγματοποιήσουν πρόοδο όλα τα κράτη-μέλη. Είπα ότι έχουμε κάποια προβλήματα και όταν που υπάρχουν συστημικά προβλήματα με το κράτο δικαίου, έχουμε προτείνει κάποια πράγματα στο νέο ε, ε, κανονισμό για τα χρηματοοικονομικά και στη νέα πρόταση που σχετίζεται με αυτό τον κανονισμό ώστε η υλοποίηση του προπολογισμού και του κράτο δικαίου να συνδέονται μεταξύ του και το κοινοβούλιο να παίζει κάποιο ρόλο εκεί. Ε, μα υποστήριξε το κοινοβούλιο και μα υποστήριξαν και αρκετά κράτη-μέλη. Δεν θέλω να πω ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με το κράτο δικαίου, αλλά όταν υπάρχει εντοπισμένο πρόβλημα, μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό πολύ γρήγορα, διότι τα κράτη-μέλη κατά το 75% του προπολογισμού σήμερα υλοποιούν τα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση όπω πρέπει. Οπότε θα πρέπει να μπορούμε να βασιστούμε στα δικαστηριά του, στου εισαγγελεί του. Γι' αυτό το λόγο έχουμε ε, καθιερώσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και μάλιστα σε στενή συνεργασία με εσά ε, και με εσά, κυρία Πρόεδρε, με τη δική σα πίεση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έγινε όσο ισχυρή θα θέλαμε, μετά από την έκβαση τη νομοθετική διαδικασία. Αλλά τώρα είναι γεγονό ε, με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών και πιστεύω ότι στο όλο συνολικό πλαίσιο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου ο Ευρωπαίο Δημόσιο Εισαγγελέα θα πρέπει να αναλαμβάνει μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο, ο οποίο να εξελιχθεί και περισσότερο στην πρακτική συνεργασία με τα κράτη-μέλη μα τα επόμενα χρόνια. Για την Τσεχική Δημοκρατία. Uh, uh, Υπάρχουν πολλά θέματα εγχώριας πολιτικής. Δεν θα σχολιάσω τώρα εδώ ο πολιτικού στην Τσεχική Δημοκρατία. Δεν είναι δικός μου ρόλος, το ρόλο της Κομισιόν. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι έχουμε λάβει την καταγγελία και δράμε όπως πρέπει. Δεν θα πω έρευνα, γιατί έρευνα είναι νομικός όρος. Δεν έχουμε φτάσει σε έρευνα, αλλά το εξετάζουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Γιατί, διότι στην Κομισιόν πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μηδενική ανοχή σε θέματα απάτη και σύγκρουση συμφερόντων σε οικονομικά ζητήματα. Το εξετάζουμε. Θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία και επειδή είναι πολιτικό το θέμα, σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να είμαστε υπερβολικά ακριβεί από νομική άποψη. Γιατί δεν θέλω να παίξω εγώ ένα πολιτικό παιχνίδι που παίζουν πάντα τα κράτη-μέλη και δεν θέλω να κρίνω οποιονδήποτε παίζει οποιοδήποτε παιχνίδι, γιατί δεν του γνωρίζω, αλλά έχουμε μια κατηγορία, έχουμε λάβει καταγγελίε και αιτήματα, το εξετάζουμε, διότι για να υπερασπίσουμε το κράτο δικαίου θα πρέπει και εμεί να συμπεριφερόμαστε βάσει του κράτου δικαίου. Οπότε και η Κομισιόν, όσο εμπλέκεται και ο Γενικό Διευθυντή μα, κ. Κόκκανη, σα εξήγησε σήμερα το απόγευμα ποιοι είναι οι κανόνε, ποιοι είναι οι νέοι κανόνε ε, βάσει του 61, ποιοι είναι οι νέοι να δούμε τι γινόταν στο παρελθόν βάσει των παλιών κανόνων, γιατί δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο κράτο δικαίου, τι γίνεται τώρα με του νέου κανόνε. Συγκεντρώνουμε τα στοιχεία και είμαστε σε στενή επαφή με τι τσεχικέ αρχέ. Και θα σα ενημερώσουμε μόλι θα έχουμε αυτά τα στοιχεία που θα μα επιτρέψουν να λάβουμε μια απόφαση, να κάνουμε μια κρίση. Την οποία θα κάνουμε μόνο εφόσον θα έχουμε όλα τα στοιχεία για αυτή, γιατί είναι η καλύτερη άμυνα για την υπεράσπιση του κράτου δικαίου. Μετά έχουμε τι ερωτήσει ε, του κ. Σα ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Αυτό που είπατε το λαμβάνουμε πολύ στα σοβαρά τελευταία χρόνια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οι ομάδε εμπειρογνωμόνων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανεί και ισορροπημένε και σε θέματα ισότητα των φύλων, ε, θέμα που ξανανέφερα προηγουμένω. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να υπερβάλλουμε για τη σπουδαιότητα των ομάδων εμπειρογνωμόνων, γιατί παρατηρώ ότι η λειτουργία τη Κομισιόν εδώ και χρόνια και μια φορά έμαθα από ένα γενικό διευθυντή ότι αν δεν θέλει να κάνει κάτι, φτιάξε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Οπότε μερικέ φορέ είναι υπερβολική η χρήση του. Αλλά τέλο πάντων, αν υπάρχουν τέτοιε ομάδε εμπειρογνωμόνων, πράγματι θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ό,τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και βάσει φίλων και βάσει συμφερόντων και να χαρακτηρίζονται από επαρκή εμπειρογνωμοσύνη ε, και προσβλέπω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Το ίδιο και για τους καταγγέλτες, τους whistleblowers. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Έχουμε κανόνες που δεν υπάρχουν στα κράτη-μέλη. το λέμε και αυτό. Οι κανονισμοί που υπάρχουν εδώ πέρα, ο εσωτερικός κανονισμός έχει κανόνες εδώ και χρόνια. Εγώ θα έλεγα ότι αυτέ είναι ακραίε περιπτώσει. Σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει τίποτα άλλο, γιατί έχουμε και άλλα μέσα. Έχουμε την υπηρεσία δημοσιολάβηση, υπάρχει δυνατότητα τη Όλαφ, του να πάει στου ανωτερού του. Θα έλεγα λοιπόν στι περισσότερε περιπτώσει έχουμε λύσει για τα προβλήματα που εντοπίζονται, αλλά συμφωνώ μαζί σα Υπάρχει και μια ανθρώπινη πλευρά. Δεν θα σχολιάσω για επιμέρου περιπτώσει γιατί δεν θα ήταν δίκαιο για κάποια άτομα αλλά ξέρω ότι έχουν μιλήσει με τον πρώτο αντιπρόεδρο για αυτό και ευχαριστώ να το συζητήσουμε μαζί ιδιωτικά οποιαδήποτε στιγμή θέλετε για να προστατεύσουμε το ιδιωτικό απόρριτο των ελλογοατόμων. Κύριε Σαλαφράγκα, ευχαριστώ και εσά ε, για την υποστήριξή σα ε, για το συνολικό αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία απαλλαγή. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το συντονισμό στον τομέα της επικοινωνίας και της διαφάνειας αυτό το θέμα απαιτεί συνεργασία μεταξύ μα πριν από τι ευρωεκλογέ. Εμεί στην Επιτροπή ω Δημόσια Υπηρεσία, εσεί ω πολιτικό θα πρέπει να μαχηθείτε. Ανέφερα κάποια παραδείγματα στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον την ιστοσελίδα ε, αποτελέσματα από τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σα καλώ να πάτε να το δείτε. Ανέφερα κάποια παραδείγματα προηγουμένω στην εισαγωγή μου για να δείτε τι ε, επιτυχάνει ο προπολογισμό στον ένα ή τον άλλο κλάδο. Α μην αφήνουμε τι εθνικέ αρχέ να λένε ναι, αυτή τη γέφυρα τη εμεί, να λένε και τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ φορέ δεν είναι μόνο γέφυρε, είναι και άλλα ε, υποδομέ υψηλή τεχνολογία. Ε, ανεμόμυλοι, ε, ανεμογεννήτριε. Ε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να τα παρουσιάσουμε με πιο φιλικό τρόπο στην ιστοσελίδα. Κάποιοι θα μας κατηγορούν για προπαγάνδα. Προπαγάνδα δεν είναι όταν λέμε τα πραγματικά στοιχεία. Εμείς απλά τα στοιχεία παρουσιάζουμε και φροντίζουμε να συμφωνούν με αυτά που έχουν γίνει πραγματικά. Το έχετε δει στην ετήσια έκθεσή μας για τη διαχείριση και την απόδοση. Υπάρχουν και στοιχεία εκεί, γιατί ξέρω ότι ε, ενδιαφέρει το θέμα και την κυρία Γιάλα. Θα δείτε εκεί κάποιους κλαδούς ε, και μπορείτε να πάρετε από εκεί δύο-τρεις προτάσεις αν σας χρησιμεύουν. Τις έχουμε βάλει εκεί ως ε, σύνοψη μαζί με όλα τα στοιχεία και τα νούμερα. Ευχαριστούμε για τα θετικά σα σχόλια για τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Για αυτή τη στιγμή για τη συμφωνία Μερκοσούρ πρέπει να σα πω ότι εργαζόμαστε σκληρά. Αλλά δεν είναι μόνο στα δικά μα χέρια, ε, εξαρτάται και από τι χώρε Μερκοσούρ που θα έλεγα η ε, Μερκοσούρ είναι πιο περίπλοκος οργανισμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είμαι βέβαιο ότι στη διάρκεια τη θητεία μα θα τα καταφέρουμε σίγουρα, όχι η Κομισιόν μόνο. Έχουμε πολλού ανθρώπου στην Κομισιόν, πολλέ υπηρεσίε που εργάζονται για αυτή τη συμφωνία και το παρακολουθώ φυσικά στενά μέσω τη Γενική Γραμματεία, Έχουμε τη DG Agri αλλά και πολλού άλλου. Όταν μιλάμε για κανονιστική συνεργασία, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη δουλειά μα για την πολυμορφία. Και οι Αμερικανοί εταίροι μα το παρακολουθούν πολύ στενά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ενώ οι ΙΠΑ αποσύρονται, εμείς πηγαίνουμε στις διάφορε περιοχές του κόσμου και μπαίνουμε εκεί. Και αυτό το μήνυμα επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πέραν των δημοσιονομικών ζητημάτων που συζητάμε. Κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα όλε τι ερωτήσει και τι δικέ σα που ήταν οι πιο δύσκολε, όπω πάντα, όπω πρέπει. Και είμαι στη διάθεσή σα ε, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση και την ανάλυση με τα επιμέρους mail εδώ ή με την Επιτροπή σα, αν το κρίνετε απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σα. Ευχαριστούμε. Θα κλείσουμε σε λίγο, αλλά δίνουμε το λόγο στον συνάδελφο Πυρίνσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια διευκρίνηση νομίζω ότι απαιτείται. Αυτό που ρώτησα εγώ είναι αν η Επιτροπή που είναι υποχρεωμένη από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, αν η Επιτροπή θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο ενημέρωση για τη διοικητική διαδικασία που ακολουθεί για το διορισμό ανωτάτων στελεχών και για τους κανόνες της διαδικασίας Στι περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή οφείλει να το κάνει, οφείλει λόγω του ψηφίσματο. Εγώ δεν έκανα ερώτηση για τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Γενικού Γραμματέα, άρα δεν καταλαβαίνω καθόλου την απάντηση που έδωσε. Ήταν μάλλον μια προσπάθεια να με μαλώσει και να απευθύνει τις ερωτήσεις προς εμένα. Ίσως λοιπόν δεν κατάλαβε αυτό που ρώτησα. Φαντάζομαι ότι νομίζει ότι δεν έχουν βάση αυτά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Οπότε θα πρέπει η Επιτροπή να μας δώσει κάποια ε, απάντηση, να μας πει ότι δεν θεωρούμε ότι πρέπει να σας δώσουμε αυτή την ενημέρωση. δεν νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας πιστεύει ότι ο ίδιος μπορεί να αποφασίζει αν ε, είναι βάσιμο το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ή όχι. Μήπως πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Μήπως πρέπει η Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό. Γιατί δεν μιλάμε για οποιασδήποτε συστάσεις, μιλάμε για συστάσεις που απευθύνονται στον πυρήνα της ακαιρεότητας της Επιτροπής. Πιστεύω λοιπόν είναι τώρα βέβαια η πρώτη φορά που συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας στη διαδικασία απαλλαγή και σιγά σιγά ίσως μάθει με το πέρασμα του χρόνου ότι δεν είναι πρέπον ένας Γενικός Γραμματέας να προσπαθήσει να συνετίσει τα μέλη της Επιτροπής μας. Θα μάθει ότι εμείς κάνουμε τις ερωτήσεις και η Επιτροπή απαντά. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Ε, υπάρχει το ψήφισμα. Να σας ρωτήσω λοιπόν πότε μπορούμε να περιμένουμε τις απαντήσεις της Επιτροπής της ε, ε, τη διαμεσολαβήτριας. Κύριε Πρόεδρε, ε, λέει ο κύριος Ζελμάγερ, ε, δεν ήθελα να στραφώ κατά του κυρίου Ευρωβουλευτού. Η Επιτροπή πάντοτε δίνει απαντήσεις και σε όλα αυτά τα θέματα θα απαντήσουμε και οι απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις ε, του διαμεσολαβητή θα απαντηθούν. Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτές τις ερωτήσεις, διότι αυτό είναι θέμα του σώματος των επιτρόπων. Όταν θέτετε ερωτήσεις σε μένα, πάντοτε ευχαρίστως απαντώ. Είμαι στη διάθεσή σας και στη διάθεση τη δική σας κύριε Πυρίνσκι. Το τι αποφασίζει τελικά να κάνει το Σώμα των Επιτρόπων είναι απάντηση των Επιτρόπων, είναι δική του απόφαση και είναι πολιτικού επίπεδου. Εμένα μπορείτε να με κρίνετε με βάση τα ε, προσωπικά μου προσόντα και όχι με βάση τις φήμες. Αυτό είπα. Κυρία Πρόεδρε, να είμαι και εγώ πολύ σύντομο να πω πως συμφωνώ με τον ε, συνάδελφο. Είναι το κοινό βούλιο που πολιτικά ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι το αντίστροφο. Αλλά δεδομένου πως αυτή η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο δέχτηκαν ένα ψήφισμα, το οποίο ήταν ad είναι σωστό για να δημιουργήσουμε μια καλή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, να τον ακούσουμε ε, ανεξάρτητα με το γεγονός πως εμείς κάνουμε τον έλεγχο σύμφωνα με το ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε και το οποίο στην παράγραφο 22 λέει η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπε πως νομικά ήταν άμεμπτη η διαδικασία, παρόλο που θα μπορούσαν κάποια στοιχεία να έχουν βελτιωθεί. Μάλιστα, κατανόησα τη διαδικασία της Επιτροπής για το, σχετικά με το ποιος ε, δίδει τις ερωτήσεις ε, στο ψήφισμα. Θα πρέπει να μας δοθεί απάντηση στο ψήφισμα. Ναι, ε, ε, ξέρουμε, θα θέλαμε να έχουμε μια απάντηση. Σας δίνουμε το λόγο για άλλη μια φορά. Είμαι 100% πεπισμένο πω οι επίτροποι θα σα απαντήσουν. Μου το είπε και ο κύριο Έτιγκερ, αλλά κατανοήστε πω εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συμμετάσχω στην ε, σχεδιασμό απαντήσεων που έχουν να κάνουν με το διορισμό μου. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά, όχι μόνο το ψήφισμα, αλλά και την συζήτηση που γίνεται μεταξύ μου Και έχετε δει και τα στοιχεία που δώσαμε για το πώ διορίζονται οι ανώτεροι υπάλληλοι, κατά τη γνώμη μα βασιζόμενοι στα προτερήματα και όχι εθνικό και κάναμε και ένα γύρο τραπέζι με τον κύριο Έτιγκερ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσει η διαδικασία και να συζητηθούν ε, και τα θέματα αυτά εν και των όσων πιστεύουν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, γιατί είναι σημαντικό. Μετά από τούτο το επεισόδιο, το οποίο Δυστυχώ έτσι συνέβη και είμαι ο πρώτο που λυπάται, γιατί εγώ υπέφερα περισσότερο από του υπόλοιπου, να προχωρήσουμε και να λειτουργεί όσο δυνατόν καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ρούσο, θέλετε να απαντήσετε. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τη συζήτηση, κατέγραψα τα θέματα αυτά. Τα λαμβάνουμε υπόψη για τις δικές μας εργασίες που τρέχουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να πω κάτι συγκεκριμένο. Frau Kollegin Ayala, bitte. Κύριε Αγιάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω πως πρέπει καταρχήν να σας ευχαριστήσω για μια συζήτηση που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και που επίσης αφήνει και κάποια έγγραφα για ανταλλαγές απόψεων και εγγράφων που θα ακολουθήσουν και που θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντα όλα αυτά και θα μας εξηγήσουν πως ο Γενικός Γραμματής κ. Σελμάγερ θεωρεί πως μπορεί να βελτιώσει κάποια από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε εδώ. Εγώ να σας πω πως θα επιστρέψω ε, μια φορά ακόμα σε ένα θέμα που για μένα είναι σημαντικό και το οποίο προέκυψε τώρα. Όταν ξεκίνησα να μιλάω είπα πως έχουμε κάποιες καταγγελίες και έχουμε και κάποιες απαντήσεις και στις απαντήσεις τις επόμενες θέλουμε να αλλάξει ο τόνος και μιλώ για την 51 όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πιστεύει πως οι διαδικασίες διορισμού των senior managers δεν είναι η κατάλληλοι. Δεν μιλώ τώρα αυτή τη στιγμή για το γενικό διευθυντή καθόλου, αλλά για άλλους ε, πολλά ήταν τα προβλήματα που συναντήθηκαν και το είπε αυτό η Επιτροπή μας, οπότε το πλαίσιο μας είπε η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή πως το πλαίσιο είναι σταθερό και επαρκές. Εδώ εμείς θα διαφωνήσουμε. Θεωρούμε πως το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνονται όλοι αυτοί οι διορισμοί χρειάζεται βελτίωση και νομίζω ότι ναι, υπέφερε ο κύριο Σελμάγερ. Αλλά έχουμε το ψήφισμα το οποίο ε, ε, τελεία τελεία και ακόμα ακόμα διαπραγματευτήκαμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων και αυτό νομίζω αποδεικνύει πως το σύστημα ως έχει δεν εξασφαλίζει ότι είναι επαρκώς σταθερό. Γιατί κάποια στιγμή κάποιος υπέστη βλάβη παρόλο που ήταν νόμιμη και αυτό που καταλάβαμε εμεί είναι ότι δεν υπήρχε καν σύστημα ή κανονισμό συγκεκριμένος για αυτό το διορισμό. Και από εκεί δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Η ερώτηση 51, λοιπόν, νομίζω εκεί η απάντηση θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Τουλάχιστον έτσι κατανοώ τα όσα μας υποσχέθηκε ο κύριος Σαλμάγερ, τον οποίο για μια φορά ακόμα καλωσορίζω. Και θεωρώ πως θα συνεργαστούμε μαζί του θαυμάσια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι ξεκινάει μια λαμπρή φιλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε για την εμβάθυνση αυτής της φιλίας. Θα σας ζητήσουμε και ένα αντίγραφο της επιστολής σας προς τη Γενική Διεύθυνση. Αυτό που αναφέρετε στην αρχή, αν μπορείτε να μας το δώσετε σε ένα αντίγραφο γιατί αυτό είναι το βασικό αντικείμενο της Επιτροπής μας. Μας ενδιαφέρει να έχουμε τα κείμενα αυτά. Στο πλαίσιο της καλής φιλίας την οποία μόλις ξεκινήσαμε θα σας δώσω αυτό το αντίγραφο, για ο κ. Ζαλμάγιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Ε, από εδώ και πέρα θα λέμε καλά Χριστούγεννα συνέχεια. Και η θερμοκρασία έχει γίνει Χριστουγεννιάτικη. Εμείς συνεχίζουμε με τα σημεία της μερίσιας διάτραξης. Περνάμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάτραξης. Μελέτη για την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα εισηγητής ο κ. Σπερίνσκι θα μας παρουσιάσουν τη μελέτη, που είναι μια μελέτη του ΣΕΠΣ. Είναι μεγάλος ο πειρασμός να εγκαταλείψει κανείς την αίθουσα, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω όσους φεύγουν να φύγουν ησύχω και ταχαίως για να συνεχίσουμε. Go ahead, please. You have the floor. Thank you very much. Okay, I can start. Um, well, I'm going to transfer you from a very exciting... Λοιπόν, θα σας μεταφέρω από μια συναρπαστική συζήτηση σε μια πιο γήινη την ε, εκ των προτέρων αρεσιμότητα των ε, ταμείων ESI. Ε Δεν είναι πολύ συναρπαστικό το θέμα, αλλά ήταν ενδιαφέρουσα η μελέτη Ονομάζομαι Χόρχε Νούνιες, ε, είμαι από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών Πολιτικής ε, και δίπλα μου είναι ο Μπέρτο Μοσμέτσο που έκανε το μεγαλύτερο κομμάτι της σκλήρης δουλειάς και την ανάλυση των δεδομένων. Όλα τα καλά στοιχεία λοιπόν είναι δικά του, αυτός τα έχει φτιάξει και τα λάθη επίσης. Σε αυτόν θα απευθυνθείτε για τεχνικές ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Εγώ θα βασιστώ στα μηνύματα που απορρέουν από αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, σε τι εστιαστήκαμε μαζί τη ΣΑΝΑ να δούμε την πρόοδο της εκπλήρωσης της αρεσιμότητας ε, ε, για τα κονδύλια ESI. Εμείς αυτό το κάναμε μέσω συνεντεύξεων με τις διαχειριστικές αρχές για να δούμε τις απόψεις τους. Δηλαδή είδαμε τα δεδομένα, δεν τα αναλύσαμε μόνο, πήγαμε και σε συνεντεύξεις. Μία από τις ερωτήσεις ήταν, ήταν χρήσιμο έχει νόημα όλο αυτό το εγχείρημα και τι σημαίνει. Ήταν αναλογικό όσον αφορά τα αποτελέσματα, άξιζε τον κόπο, ήταν υπερβολικά βαρύ. Ποια ήταν η σχέση κόστους-οφέλους. Και τέλος, υπάρχουν κάποια διδάγματα για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, για τον επόμενο κανονισμό κοινών διατάξεων, όπου δεν θα ονομάζονται εκ των προτέρων αρεσιμότητα, αλλά προϋποθέσεις ε, δράσης. Ε, ο κανονισμός των κοινών διατάξεων όπως διατυπώνεται, διατυπώνει τις διατάξεις για την εξάντε αιρεσιμότητα. Εκεί υπάρχει ένας ορισμός που έχω βάλει εδώ στην οθόνη. Αξίζει να δει κανείς τις ελάχιστες απαιτήσει για να υπάρχει πραγματική αποτελεσματικότητα και για να είναι η δαπάνη των ε, κονδυλίων αποτελεσματική. Εδώ μιλάμε για υλοποίηση οδηγιών που σχετίζονται άμεσα ε, με κάποιου τομεί ε, παρέμβαση. Δεν μπορεί δηλαδή κανεί να πάρει χρήματα για να φτιάξει ένα εργοστάσιο καθαρισμού υδάτων, αν η οδηγία για την επεξεργασία των λιμάτων δεν έχει υλοποιηθεί σε μια χώρα. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή το νομοθέτημα. Δηλαδή ουσιαστικά αν δεν υπάρχει το κεκτημένο δεν σας χρηματοδοτούμε. Αυτό είναι κάπου το μήνυμα. Παρότι το λέμε ήπια, γιατί υπάρχει κάποιος χρόνος, αλλά αυτή είναι η τελική, το τελικό σκεπτικό. Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χρηματοδοτεί κάτι για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμα κανόνες. Η εκ των προτέρων αρεσιμότητα λοιπόν ενισχύει τι δυνατότητε υλοποίηση και νομική συμμόρφωση βοηθά. Υπό την έννοια ότι ζητά από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τις ε, ικανότητες και τις δυνατότητες ε, για συμμόρφωση με οδηγίες και κανονισμούς. Υπό τον όρο όμως, ε, επειδή μιλάμε για διαρθρωτικά ταμεία, δεν έχουμε διαδικασία παραβάση εδώ από τις Γενικές Διευθύνσεις, ουσιαστικά υπό τον όρο ότι το κράτος μέλος ζητά ευρωπαϊκά κονδύλια. Εάν απλά υλοποιεί κάποιο τι οδηγίε δεν είναι περιφερειακή πολιτική. Αυτό πρέπει να έχει να κάνει με τι σχετικέ αρχέ. Το θέμα εδώ είναι να δούμε πώ δαπανώνται κάποια κονδύλια. Ε, όταν λαμβάνει κανεί ενίξη, πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση. Η συμμόρφωση πρέπει να υπάρχει ούτω ή άλλω, αλλά τότε η διαδικασία είναι διαφορετική. Υπάρχουν 48 εξάντε ερεσιμότητες, 7 ε, γενικέ 29 θεματικέ, 12 ε, αφορούν συγκεκριμένα ταμεία. από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας. Ε, εκεί έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, ρεσιμότητες εκ των προτέρων. Η διαδικασία, όπως εφαρμόστηκε, είχε ως εξής οι χώρες, πρώτα απ' όλα, αφού έχουν έτοιμο το πλαίσιο υποστήριξη, υπογράφουν μια συμφωνία εταιρική σχέση με την Κομισιόν. Εκεί υπάρχει συμφωνία για τη γενική στρατηγική. Βάσει αυτής της συμφωνίας δημιουργούνται τα επιχειρησιακά προγράμματα με τις προτεραιότητες δράσεις ανατομέα τα ποσά και μετά από αυτό ανάλογα με το ποιες θα είναι οι δράσεις θα πρέπει να εκπληρούνται οι εκ των προτέρων ερεσιμότητε. Ε, και η έννοια του εκ των προτέρων σημαίνει σε έναν ιδανικό κόσμο ότι οι προποθέσει πρέπει να πληρούνται πριν ξεκινήσει η προγραμματική περίοδο. αλλά επειδή πάντα καθυστερεί η προγραμματική περίοδος ε, ότι δεν ε, έχουμε πρόγραμμα να το ετοιμάσουμε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση γι' αυτό. Τι γίνεται λοιπόν ε, στην πράξη για να σας δώσω μια εικόνα οι γενικές αιρεσιμότητες θα τις δούμε αργότερα εκεί είχαμε το 61% των, όπου οι αιρεσιμότητες πληρώνονταν στα κράτη-μέλη το 39% όχι και για τους θεματικούς στόχους ήταν το ίδιο 63. Δηλαδή σχεδόν το 40% των ε, εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων δεν εκπληρούνταν έγκαιρα στην Ευρώπη γενικότερα. Όταν δεν υπάρχει αυτή η εκπλήρωση, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εκπονήσουν σχέδια δράσης ε, για την εκπλήρωση. Τα σχέδια δράσης αυτά θα παρακολουθούνται στη συνέχεια και υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για τις χώρες εντό των οποίων οι χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά τα σχέδια δράση. Πώς ε, είχε η κατάσταση, τα έγγραφα τα... μας ήρθαν μέχρι το Μάρτιο του 2018 και ξέρω ότι εμφανίστηκε και ένα νέο έγγραφο μετά από την έκθεση αυτή, αλλά λείπει κάτι δηλαδή, αλλά θα το προσθέσω. Είχαμε 1.401 σχέδια δράση σε όλου ε, τι θεματικέ και γενικέ εκ των προτέρων ερεσιμότητε. Αυτό έχει να κάνει με διάφορε αρχέ. Ποιε αρχέ, ανάλογα με το πώ είναι δομημένες και οργανωμένε οι χώρε. Η αρμόδια διαχειριστική αρχή είναι αυτή εδώ. Άλλε έχουν πολλέ, άλλε έχουν λιγότερε. Αυτό έχει να κάνει με τι εσωτερικέ διοικητικέ δομέ παρά με οτιδήποτε άλλο. Οπότε σε κάποιε χώρε είναι ελάχιστε, αλλού πολλέ παρόμοιου μεγέθου εξαρτάται από την ε, κυβερνητική δομή ουσιαστικά, από την κυβερνητική δομή κάθε χώρα. Κάθε χώρας. Εδώ έχουμε τον κατάλογο και θα βρείτε γενικά ζητήματα όπως δημοσίες συμβάσεις, ε, την ισότητα των φύλων, τους ε, κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Αφορούν όλα τα προγράμματα. Έχουμε μετά τα θεματικά, τις θεματικές ρεσιμότητες που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Πάμε να δούμε την κατανομή. Ε, στην αρχή τα μπλε κουτάκια είναι οι κεντρικές και ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπετε έχουν να κληρώσουν πολλές αιρεσιμότητες σε σύγκριση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Και περισσότερο από τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι γιατί είναι μεγάλη, οι περισσότεροι δικαιούχοι κονδυλίων εκεί και υπάρχει και μια σχέση φυσικά μεταξύ της ε, κατάταξης και των τομέων που λαμβάνει υποστήριξη. Αν προκτήκα μια χώρα σε φάση σύγκλησης, ε, η περιοχή οι χώρε λοιπόν που λαμβάνουν λιγότερα κονδύλια θα έχουν λιγότερα τέτοια σχέδια δράση. Οι παλιότερε χώρε επίση έχουν λιγότερα τέτοια γιατί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία όσον αφορά την υλοποίηση στι περισσότερε περιπτώσει. Αλλά όχι πάντα. Αυτό το ανέφερα ήδη στην εικόνα, οπότε μπορούμε να το περάσουμε. Οι διοικητικέ δομέ παίζουν ένα ρόλο και εδώ μπορούμε να δούμε την κατάσταση εκπλήρωση ανά χώρα. Παρατηρούμε ότι στι περισσότερες χώρες οι περισσότερες έχουν εκπληρώσει τα σχέδια δράση έγκαιρα. Και εδώ βλέπετε τα σχέδια δράση αναχώρα. Το πρώτο που βρήκα ενδιαφέρον σε αυτή τη μελέτη ήταν αυτό. Και μου φάνηκε και λίγο περίεργο. Αν πάμε να δούμε χώρες μεγέθους Ισπανίας, είχε 32. Οι αυτόνομε περιφέρειες επίσης υπήρχαν της Ισπανίας, αλλά με πολύ σαφή δομή αρμοδιοτήτων και κατανομή εξουσιών. Οπότε τα Υπουργεία εδώ ε, λειτουργούν συντονιστικά με πολύ σαφή τρόπο. Η Ισπανία λοιπόν είχε 32. Η Ισπανία παρουσιάζει υψηλή συμμόρφωση. Σε ελάχιστο τομεί είχαν πρόβλημα συμμόρφωση ε, με τα σχέδια δράση. Ε, ενώ στην Ιταλία είναι 319. 320 γιατί το ένα δεν εκπληρώθηκε. Το ζήτημα λοιπόν, το ερώτημα ήταν γιατί. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μάθαμε από τη συνέντευξη ότι αυτό οφείλεται στι κρατικέ δομέ. Πολλέ διαφορετικέ αρχέ ε, ταυτόχρονα αρμόδιε για παρόμοια πράγματα. Επανάληψη καθηκόντων, διπλασιασμό καθηκόντων, πολύ δύσκολη διακυβέρνηση. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ ενδιαφέρον όπω προκύπτει από τι εκ των προτέρων αρεσιμότητε. Μας βοηθούν να ανακαλύψουμε πόσο ε, συγκεντρωμένη είναι η διακυβέρνηση σε κάποιες χώρε και πόσο καλό συντονισμό υπάρχει. Θα σα εξηγήσω αργότερα ποια ήταν η δική του άποψη για αυτό το εγχείρημα. Ε, σε μια χώρα όπω η Ιταλία κάναμε πολλή δουλειά και η Ελλάδα επίση είναι ενδιαφέρουσα όσον αφορά δεδομένο το μέγεθό τη και η Πολωνία δείχνει, έχει κάποιο ενδιαφέρον ε, για το πώ συντονίζει τα πράγματα και η κεντρική κυβέρνηση και μην ξεχνάμε ότι όσο περισσότερα χρήματα παίρνει κανεί, τόσο περισσότερα σχέδια δράση πιθανότητα πρέπει να εκτελέσει. Κάτι που θέλω να προσθέσω σε αυτή την εικόνα είναι ότι στην τελευταία έκθεση δραστηριοτήτων είχαμε μία αναστολή. Και τρεις περιπτώσεις όπου δεν καταφέραν να, διαχειριστούν τα σχέδια δράσης. Αλλά είναι 95% ουσιαστικά η εκπλήρωση. Είναι πολύ καλό. Αλλά στην έκθεση δεν καθορίζεται πού έγιναν αυτές οι αναστολές. Εγώ δεν τις είδα. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι πόσο αυτό το εγχείρημα επηρέασε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα ποιο ήταν το κόστος όλων αυτών του να εξετάσουμε ολόκληρη την νομοθεσία, του να μπορείς κανείς να ακολουθήσει, να εφαρμόσει όλη την νομοθεσία για να λάβει τα κονδύλια. Είδαμε μια διαφάνεια Όπω βλέπουμε στη διαφάνεια αυτή ε, εξαρτάται από, τις, ε, από τα μεγέθη. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι οι περιφέρειες που είχαν σχέδια δράση. και που δεν συμμορφώνονταν με τα εξάντια, είχαν χαμηλότερο ποσοστό εκπλήρωσης, χαμηλότερο ποσοστό απορρόφησης. Όταν έχει κάνει μια προγραμματική περίοδο που αρχίζει καθυστερημένα, και όταν υπάρχουν πολλοί άλλοι συντελεστέ που επηρεάζουν τα πράγματα, αλλαγέ στου κανονισμού, είναι δύσκολο να ξέρει κανεί καθαρά ότι φταίει η εκ των προτέρων αρεσιμότητα για την καθυστέρηση. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανεί τη σύνδεση. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, εμεί ε, κάναμε μια έρευνα ε, η οποία είπε ότι μόνο το 10% συμφωνεί ότι επηρεάζεται αρνητικά η απορρόφηση, η υλοποίηση δηλαδή. 38% συμφώνησαν, αλλά το 10% διαφωνούν. Και 42% ήταν αναποφάσιστοι. Δεν είπα δηλαδή οι περισσότερες αρχές ότι αυτό επηρέασε τα πράγματα. Πιστεύω όμως ότι οι περισσότεροι το αισθάνθηκαν. Now, which were another question we were μια άλλη ερώτηση που τέθηκε ήταν ποια ήταν τα σημαντικότερα. Αυτοί που θεώρησαν ότι αυτά ήταν πολύ σημαντικά ήταν οι αιρεσιμότητες για την κρατική ενίσχυση, δηλαδή πώς θα υπάρχει συμμόρφωση με τους κρατικούς κανόνες ε, θεώρησαν ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό και ότι ήταν κρίσιμη σημασία και οι δημόσιε συμβάσει επίση. Και τα δύο αυτά εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από την ερεσιμότητα. Και εκεί υπήρχαν τα περισσότερα προβλήματα, ενώ για άλλα πράγματα είπαν ναι, χρειάζεται κάποια μικρό προσαρμογή, αλλά όχι το ίδιο βάρος. Αλλά ε, αυτά ήταν τα γενικά για τα θεματικές, ε, η διαβίου μάθηση, τα σχέδια μεταφορών. Αυτά είναι στρατηγικές οι προετοιμασίε, για στρατηγικές, οι απαιτήσει. Ε, στους τομείς των μεταφορών της διαβιομάθησης, της καινοτομίας, της έρευνας. Εκεί θεωρούνται οι πολύ σημαντικές και επηρέασαν τη βελτίωση. Και αυτό μας λένε ότι επηρεάζουν τη βελτίωση των στρατηγικών. Κάναμε μελέτες περιπτώσεων στις χώρες αυτές, Βουλγαρία, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία. Ζητήσαμε τις απόψεις τους με άμεσες συνεντεύξεις με απευθεία συνεντεύξει. Επιπλέον, διότι έγινε η έρευνα σε όλη την Ευρώπη με όλες τις διαχειριστικέ αρχές, αλλά μετά κάναμε και τηλεφωνικές συνεντεύξει ε, σε διάφορες χώρες. Συνολικά πρέπει να πω ότι οι περισσότερες χώρες ήταν πολύ πιο θετικές ε, για τι εκ των προτερνερισμότητες από ό,τι περίμενα και εγώ ίδιο. Γιατί, διότι σε ένα πράγμα είχα δίκιο. στι περισσότερε περιπτώσεις θεωρούσαν ότι η προετοιμασία για τη συμμόρφωση με τι εκ των προτέρων πήγε μια χαρά. Αλλά εκεί όπου υπήρξαν τα περισσότερα προβλήματα είχαμε και την πιο θετική αντιμετώπιση. Εκεί που ε, δυσκολεύτηκαν περισσότερο ε, ε, ήταν και δύσκολο να μας προσθέσουν ποιο ήταν το πρόβλημα. Ήταν αυτοί που δυσκολεύτηκαν να υλοποιήσουν τα συστήματα. Οι χώρες φυσικά που τα κατάφεραν μια χαρά θεώρησαν ότι ήταν επαχθείς ε, και χωρίς ε, κανένα αποτέλεσμα το όλο αυτό το εγχείρημα. Γιατί, διότι όταν κάποιος ήδη συμμορφώνεται ας πούμε με την οδηγία για τα ύδατα, το γεγονός ότι υπάρχει αιρεσιμότητα εκ των προτέρων που απαιτεί να δείξει στην DG Regio ότι συμμορφώνεσαι ενώ η Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο θα πρέπει να γνωρίζει ήδη ότι συμμορφώνεσαι, αυτό τους ήταν... Τους δημιουργήσε και έκπληξη και τους δημιουργήσε και πολύ κόπο γιατί το, οι αρμόδιοι δεν ήταν και υπεύθυνοι και για τα περιβαλλοντικά θέματα και το, μας έλεγαν το, ότι το να απαιτήσουμε τώρα από αυτούς να αποδείξουν στην Κομισιόν ότι υλοποιούσε κάτι καλά ένα άλλο Υπουργείο αυτό τους δημιούργησε λίγο κάποια δυσαρέσκεια και επίσης ήταν και δύσκολο διότι κανείς δεν καταλάβαινε το λόγο για, για τον οποίο γίνονταν τα πράγματα έτσι τα βασικά μηνύματα όμως ε, είναι τα εξής θεωρήθηκαν χρήσιμες ε, οι εκ των προτέρων σε ε, ε, χώρες που έχουν προβλήματα διοικητικών δυνατοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ειδικότερα σε μία ε, περίπτωση με, για θέματα καινοτομία θεωρήθηκε ότι ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις. Απαιτεί το κάποια στρατηγική στο πλαίσιο τη εκ των προτέρων αρεσιμότητα που έδωσε τη δυνατότητα στις αρχές να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις για να προβούν στι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Έτσι λοιπόν, όπως είπα, ήδη ήταν επαχθή. Αναφέρθηκε πολλά η περιφερική πολιτική, το είπα και εγώ. Είναι περίεργο που η περιφερική πολιτική ασκεί πίεση για την υλοποίηση πολιτικών άλλων αρχών. Και η ερώτηση εκεί έλεγε υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε διαδικασία επί παραβάση. Και εμείς είπαμε αντί να ξεκινήσουμε τη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε την περιφερειακή πολιτική για να τους οθήσουμε να κάνουν κάτι τέτοιο χωρίς να πάρουν από νομική διαδικασία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ορισμένε από τις αρχές ε, θεώρησαν ότι δεν ήταν δίκαιο να θεωρηθούν υπεύθυνε για την υλοποίηση αυτών των κανόνων από άλλα Υπουργεία. Κάτι άλλο που υπόθηκε ήταν η υλοποίηση, η επίσημη παρακολούθηση και η υλοποίηση. Έλειπε. Οι κανόνες ε, ήταν ασαφείς, ήταν πάρα πολλοί κανόνες. Οι κατευθυντήρε γραμμέ τη Κομισιόν ήταν πολλέ ε, και πολύ λεπτομερεί. Και τα κράτη-μέλη έπρεπε να αποφασίσουν πώ θα αποδείκνυαν τη συμμόρφωσή του. Το τι έπρεπε να απαντήσουν και τι τα αφορούσε ε, στι κατευθυντήρε γραμμέ ήταν δύσκολο. Σε συνέντευξη στην Ισπανία μάθαμε ότι μα είπαν ακολουθούμε όλε τι κατευθυντήρε γραμμέ γιατί δεν ξέρουμε πώ θα μα απαντήσει η Κομισιόν μετά. Και εμεί του είπαμε και και μετά τι θα γίνει να πούμε εμεί ότι θεωρούμε ότι αυτό δεν μα αφορά, αλλά μετά η Κομισιόν θεωρεί ότι μα αφορά και μα δημιουργήσει προβλήματα. Οπότε καλύτερα να απαντήσουμε στα πάντα για να τι δεν ήταν σαφέ. Η αλήθεια είναι ότι αυτέ οι εκ των πρώτων ερεσιμότητε ήταν κάτι το καινούριο και η όλη διαδικασία υλοποίηση έγινε κάπως τροχάδιν. Δηλαδή και οι δύο πλευρέ το μάθαιναν κάνοντα το, το, το, πώ γίνεται η εκ των προτέρων Ούτε για την Κομισιόν ήταν σαφέ τι είναι, ούτε η άλλη πλευρά ήξερε ακριβώ θέλαμε, θέλουν απλά και δύο πλευρέ να υπάρχει συμμόρφωση. Η Κομισιόν παρέχει βοήθεια, όλοι το συμφώνησαν σε αυτό, όλες οι αρχές κατάλαβαν ότι επρόκειτο για το καλό και των δύο πλευρών ε, να συνεργαστούν, ε, να καταφέρουν να φέρουν αποτέλεσμα. Δεν ήταν μονόδρομη επικοινωνία. Όλες λοιπόν οι αρχές ε, έμειναν πολύ ικανοποιημένε με τη στάση τη Κομισιόν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είπαν ότι ήταν επαχθέ, ε, άχρηστο και δεν του άρεσε. Παρ' όλα αυτά είπαν ότι του βοήθησε η Κομισιόν πολύ. Και συμφώνησαν. Και ευχαρίστησαν την Κομισιόν για όλα αυτά. Και οι πληροφορίες που συλλέξαμε θα μας βοηθήσουν να οργανώσουμε την επόμενη, τον επόμενο γύρο. Ο επόμενος κανονισμός ε, θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά μηνύματα από το όλο εγχείρημα. Αυτές οι υποστηρικτικές συνθήκες, τα enabling conditions και το γεγονός ότι υπήρχαν και προθεσμίες. Αυτή η διαδικασία θεωρήθηκε ότι ήταν λίγο αυστηρή αυτή η διαδικασία των εκ των προτερών και συχνά δεν ήταν πολύ προσαρμοσμένη στι πραγματικέ συνθήκε. Έβλεπα δηλαδή θετικά τι προτάσει, τι ιδέε, Ε, τους άρεσε που δεν υπήρχε χρονική δέσμευση. Έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο δράση, ε, το οποίο φτιάχνει εσύ και μετά απλά η Κομισιόν παρακολουθεί την υλοποίηση κατά τη διάρκεια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και λαμβάνει κανείς χρηματοδότηση όσο καιρό ε, ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης. Ωστόσο η παρακολούθησή του ανησύχησε γιατί Κάποια κείμενα στις μελλοντικές προτάσεις είναι σαφή. Δεν μας λένε καθαρά πώς θα παρακολουθούνται αυτές ε, οι συνθήκες, οι enabling conditions. Λέγεται ότι η Κομισιόν θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την υλοποίηση αυτών των συνθήκων και ανησυχούν ότι αυτό θα είναι πολύ γραφειοκρατικό και πολύ αυστηρό. Εμείς έχουμε να σας πούμε ότι στην πραγματικότητα Μάλιστα, η υλοποίηση κάποιου σχεδίου πρέπει να αλλάξει, να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες, όχι για να αλλάξει ο στόχος, απλά κάποια πράγματα, αν τα ακολουθεί κανείς πολύ αυστηρά, αυτό μπορεί να μην φέρνει αποτέλεσμα. Οπότε... Αυτό λίγο ανησυχεί τον κόσμο. Είναι και μια προειδοποίηση. Ουσιαστικά αυτό τι μα λένε να μην είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Μα παρακολουθείτε υπερβολικά αυστηρά. Αφήστε μα να είμαστε λίγο ευέλικτοι στην πράξη. Επίση, είπαν ότι ήταν πάρα πολλέ οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητε και οι θεματικέ αιρεσιμότητε. Εγώ θα έλεγα από την άλλη πλευρά ότι δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που κάναμε αυτό το εγχείρημα, ελπίζω ότι στο επόμενο πλαίσιο θα υπάρχουν πολύ λιγότερα να γίνουν. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι τη οδηγία θα έχει υλοποιηθεί χάρη σε αυτή την άσκηση ε, τη εκ των προτέρων ερεσιμότητα, Αλλά για να θα μας βοηθήσει να το περιορίσουμε λίγο. Ένα από τα ισχυρά μηνύματα ήταν, μας έλεγαν παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις εξάντια ερεσιμότητες ως ε, εργαλείο ε, για νομοθέτηση. Εάν μια οδηγία δεν έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μην χρησιμοποιείτε τα διαρθρωτικά ταμεία για να αποφύγετε ε, διαδικές επιπαραβάση. Αυτό ήταν ένα χειρό Το δεύτερο ήταν η αποφυγή των διαφόρων επιπέδων γραφειοκρατίας. Εγώ ο ίδιος ασχολούμαι με τα διαρθρωτικά ταμεία χρόνια. Ακόμα δεν έχω καταλάβει με τι εκ των προτέρων αρισμότητε ή του αναγκαίου όρου, του αναγκαίου πρόσφορου όρου, τα enabling conditions, πώ μπορεί κανεί να αποφύγει πέραν τη αξιολόγηση και τη παρακολούθηση των προγραμμάτων, πώ μπορεί να αποφύγει κανεί. Ε, προβλήματα με την παρακολούθηση των αναγκαίων προσφορών όρων, γιατί αυτό είναι το τελευταίο βήμα για τον έλεγχο Καλό θα ήταν να αποφεύγουμε παράλληλες διαδικασίες ή διπλασιασμό των ε, ε, γραφειοκρατικών διαδικασιών σε δύο διαδικασίες να έχουμε, δηλαδή την παρακολουθήση του επιχειρησιακού προγράμματος και από την άλλη και των αναγκαίων πρόσφορων όρων ε, της εξαντερεσιμότητας που ουσιαστικά καλύπτουν τα ίδια, στρατηγική δηλαδή. Και είχαμε και ένα σχόλιο που μας είπαν, θεώρησαν ότι η ευθυγράμμιση της εκ των προτέρων σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ήταν η ίδια με τις απαιτήσει στρατηγικού σχεδιασμού για την καινοτομία, για τα σχέδια καινοτομία, ε, για τη στρατηγική. Έχουν μια στρατηγική και μια συμφωνία εταιρική σχέση και οι εξάντε μερικέ φορέ δεν ευθυγραμμίζονταν αρκετά και μα είπαν ουσιαστικά να αποφεύγουμε διπλασιασμό των εργασιών. Επικάλυψη των εργασιών. Αυτά είναι όλα τα μηνύματα από πλευρά μου. Είμαι όλο αυτιά αν έχετε ερωτήσεις. Δεν ξέρω και ο μου δεν έχει να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Είναι ήδη ε, παρά 20. Κύριε Πυρίνσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεδομένου του ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε, θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Να σας πω καταρχήν πως καλώ τους συναδέλφους και τις επιτροπές να κοιτάξουν τη μελέτη αυτή στα πλαίσια της αξιολόγησης ε, της ενδιάμεσης αξιολόγησης που θα γίνει του χρώμου γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα κληθεί να απαντήσει στο εξής ερώτημα Πώς θα πρέπει λοιπόν αυτές οι αιρεσιμότητες, για να τις χαρακτηρίσω έτσι, θα, με τη νέα τους μορφή θα βελτιώσουν την προληπτική ρεσιμότητα γιατί βέβαια αυτή είχε κάποιο ιδιαίτερο, ιδιαίτερη δυσκολία τη στιγμή της πρακτικής εφαρμογής και πολλοί δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακριβώς πώς να συμμορφωθούν με αυτές. Και αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις σε πολλές περιπτώσεις. Τη στιγμή της απορρόφησης και χρήσης των ταμείων. Οπότε εκεί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε αυτές τις περιπτώσεις όπου είχαμε κάποιο είδους αυτολογοκρισία, δηλαδή τα κράτη-μέλη δεν καταθέτουν αίτημα ε, πληρωμής γιατί θεωρούν ότι ενδεχομένως θα τους επιβληθούν και κάποιες κυρώσεις. Και πρέπει να σας πω πως αυτά είναι αρνητικά στοιχεία που έχουμε με τη χρήση των ε, προληπτικών ερεσιμοτήτων. Όπως είπαν και αυτοί που ετοίμασαν την ε, μελέτη, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς εάν έχουμε μία διαφορά μεταξύ των όσων εφάρμοσαν το εξάντε, ε, γιατί είναι πάρα πολλοί οι διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν. Από τη μελέτη είναι σαφές πως υπάρχουν θετικά στοιχεία. Για παράδειγμα, το ότι γίνονται πιο πολλές μεταρρυθμίσεις και βέβαια η αναβάθμιση που είναι απαραίτητη για τα συστήματα στα κράτη-μέλη. Στο σημείο αυτό θα τονίσω όσα είπαν οι προηγούμενοι πως ήταν η καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω αυτό να μην έχει να κάνει με το ότι τα κράτη-μέλη ε, είναι πολύ προσεκτικά όταν σχολιάζουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην έχουν προβλήματα, αλλά θεωρώ πως ήταν η πικοδομητική αυτή η σχέση, αλλά θέλω να απευθύνω κάποιες ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να σας καθυστερώ. Για παράδειγμα, αυτά τα είδη ε, εκ των προτέρων ερεσιμότητας, την γενική και την ε, ε, εκτομιακή. Ποιες είναι, από αυτές είναι η άμεση ευθύνη της DG Regio και έχουν να κάνουν με την απόδοση και την αξιολόγηση απόδοσης αυτών των ταμείων και πώς σχετίζονται άμεσα με την ε, πολιτικής συνοχής. Και θα ήθελα να ξέρω πόσο βάρος ήταν αυτή για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρακολούθηση και αξιολόγηση ε, της συμμόρφωσης με την προληπτική ρεσιμότητα, γιατί καταλαβαίνω πως υπάρχει αυτή η δυσκολία του να παρακολουθείς πάνω από 2.000 περίπου σχέδια δράσης. Και επίση, ποια ήταν τα διδάγματα από την διαδικασία αυτή. Πώς προβλέπετε να τα χρησιμοποιήσετε τα διδάγματα αυτά για την επόμενη περίοδο. Και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την έλλειψη σαφήνειας σε κάποια από τα κείμενα που έχουν προταθεί από τον κανονισμό με τις κοινέ διατάξεις γιατί ξέρω πως αυτό δημιουργεί δυσκολίες για τα κράτη-μέλη και έχει καταγραφεί και στην ίδια τη μελέτη. Νομίζω πως όλα αυτά χρήζουν ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα ζητήσω τα δικά σας συμπεράσματα, τα έχουμε δει στην οθόνη, είναι και πολύ ε, συγκεκριμένα και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, πλήρως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ συναρπαστικά ήταν τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε. Δεν είμαι σίγουρη για την κατεύθυνση των συμπερασμάτων. Πάντως η συλλογή δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική. Από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υποθέσεων, ο κύριος Γκραντ είναι παρόν. Παρακαλώ, πείτε μας το όνομά σας. Γιολάντα Σπακόμφσκα, λέγομαι πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση Regio, δεν, δεν μπορούσε να έρθει ο κύριος Γκραντ σήμερα. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για πρώτη φορά παρουσιάστηκε σε αυτή την προγραμματική περίοδο και όπως αναφέρθηκε και για την Επιτροπή και για τα κράτη-μέλη και για τις περιφέρειες ήταν μια διαδικασία στην οποία ε, μάθαμε σιγά-σιγά. Η μελέτη τονίζει τα θετικά αποτελέσματα και χαίρομαι γι' αυτό. Οι διαχειριστικές αρχές στις απαντήσεις τους δείχνουν ότι υπήρχε θετικός αντίκτυπος παρά τον διοικητικό φόρτο. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν ε, σαφή στοιχεία για την ε, υψηλή απορρόφηση και τον αντίκτυπο των ε, των προτέρων ερεσιμοτήτων. σχολιάζοντας ένα από τα συμπεράσματά σας ότι εκ των προτέρων είχαν ως στόχο τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες, θέλω να πω το εξής. Ο στόχος των εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων ήταν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των ταμείων. Αυτό ήταν ο στόχος που είχαμε δηλώσει καταρχήν είναι σημαντικό να υπάρχει η σύνδεση με την Ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως και η οθέτηση των οδηγιών. Ε, τέθηκε το θέμα της παρακολούθησης για την επόμενη, για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ένα από τα μειονεκτήματα του τωρινού κανονισμού, όπως είπατε και εσείς, είναι ότι η Επιτροπή δεν έχει μηχανισμό παρακολούθησης της υλοποίησης των σχεδίων δράσης και παρακολούθησης του αν υπάρχει σύνδεση των στρατηγικών που με μεγάλο κόπο εγκαθιδρύθηκαν ε, και της ε, επιλογής των έργων. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο λοιπόν ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ε, την υλοποίηση εξουσιοδοτικών δράσεων σε όλη την προγραμματική περίοδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ζητάμε συνεχώς εκθέσεις για την τρέχουσα κατάσταση κάθε στρατηγικής, ούτε ζητάμε κάθε φορά ε, να ελέγξουμε τις χιλιάδες εγγράφων ε, για όλα τα προϊόντα που παράγονται από τα κράτη-μέλη κατά μία προγραμματική περίοδο, όπως είπατε και εσείς εξάλλου αυτό το οποίο υποστηρίζουμε είναι να υπάρχει κατάλληλη προσαρμογή των στρατηγικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες οι οποίες μεταβάλλονται και δεν θα είμαστε άκαμπτοι σε αυτό το τομέα. Θέλουμε όμως να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις και ότι υπάρχουν ε, οι εκ των προτέρων ερεσιμότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ακόμη και όταν αλλάζουν οι συνθήκες, οι όροι θα πρέπει να πληρούνται. Δεν θα παρεμβαίνουμε όμως εμείς στο πώς υλοποιείται μια στρατηγική. Ε, ούτε στον τρόπο προετοιμασίας της στρατηγικής, γιατί αυτό δεν είναι στις δικές μας αρμοδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό η δική μας αρμοδιότητα είναι να ελέγξουμε ε, αν συνεχίζουν ε, να υλοποιούνται, να εφαρμόζονται τα κριτήρια τα οποία έχουμε θέσει εμείς στο πλαίσιο της αιρεσιμότητας. Έγινε και μια ερώτηση για το αν η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο έχει ε, την ικανότητα να αξιολογεί το αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις. Η διαδικασία την οποία θεσπίσαμε ήταν ότι η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο ήταν υπεύθυνη για την ε, αξιολόγηση, τη διαχείριση της αξιολόγησης και υπάρχουν οι αρμόδιες ε, γενικές διευθύνσεις γιατί όπως ξέρετε η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο χρηματοδοτεί πολλούς τομείς σε όλα τα κράτη-μέλη και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ειδικοί σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων ή μεταφορών ή όλων των άλλων τομέων. Επομένως, σε συνεργασία με άλλες γενικές διευθύνσεις έγινε η αξιολόγηση. Πάντοτε όμως εξετάζουμε τη σύνδεση που υπάρχει με τη δική μας χρηματοδότηση. Η έννοια της εκ των προτέρων ερεσιμότητας είναι το να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση. Εξετάζουμε λοιπόν τα συγκεκριμένα κριτήρια και σε αυτή την προγραμματική περίοδο είχαν προσαρμοστεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα συνδέονται ακόμη πιο στενά με, τους, ε, με τις περιοχές παρέμβασης με τρόπο στο δυνατόν περισσότερο συγκεκριμένο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η μελέτη αυτή ε, φαίνεται ενδιαφέρουσα. Μας δίνει ιδέες και για την επόμενη προγραμματική περίοδο και είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια κράτη-μέλη και ποιες περιφέρειες αντιμετώπισαν περισσότερα περιστατικά εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που δεν τηρήθηκαν. Η ευθύνη ε, εκπλήρωση των προποθέσεων δεν είναι πάντοτε αρμοδιότητα των αρμόδιων υπουργείων. Στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει η αρμοδιότητα σε περιφερειακό επίπεδο και πολλές φορές υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα. και αυτό πολλές φορές κατέληξε στο να έχουμε πολλά σχέδια δράσης. Υπήρχαν δηλαδή αρμοδιότητες σε διάφορα επίπεδα και γι' αυτό χρειάστηκε να προετοιμαστούν και πολλά έγγραφα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, αν έχει κάποιος κάποια παρέμβαση, παρακαλώ. Νομίζω πως θα συμφωνήσω. Αυτό που κάνουμε είναι να παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα ε, που ουσιαστικά απηχούν τις ανησυχίες των όσων ερωτήθηκαν. Και οι προτάσεις για την επόμενη περίοδο είναι προτάσεις απλώς. Και βεβαίως οι διαχειριστικές αρχές ανησυχούν για το πώς οι προτάσεις αυτές θα εφαρμοστούν. Τι θα γίνει στο τέλος. Οπότε, επαναλαμβάνω, πρόκειται κυρίως για ανησυχίες. Δεν έχω προσωπική άποψη. Δεν έχουμε προσθέσει κάτι σε αυτή τη μελέτη, κάτι δικό μας, βασιζόμαστε στα δεδομένα που έχουμε και αν υπάρχουν κάποια σφάλματα, ε, εντάξει. Έχουμε κάποιες ε, ανησυχίες και φόβους που εκφράστηκαν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Άρα ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της μερικής διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά και περνάμε στο σημείο 21 της ημερήσιας διάταξης η γνώμη του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο 2020. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Φιγκουερέιντο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το γεγονός πως κάλεσε το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει αυτήν την παρουσίαση της γνωμοδότησής του ε, και πρέπει να σας πω πως εμείς πάντα χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε και σας κάνουμε αυτές τις παρουσιάσεις και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για συζήτηση αυτών και βέβαια και, και τη συγκεκριμένη γνώμη. Δεύτερον, στο ελεγκτικό συνέδριο αναγνωρίζουμε πως ο σχεδιασμός της ΚΑΠ Είναι εξαιρετικά περίπλοκο θέμα. Και θα έλεγα πως τα έγγραφα αυτά, τα οποία χρησιμοποιήσαμε για τα σχέδια κανονισμών που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επίσης κείμενα ιδιαίτερα περίπλοκα και θα τολμούσα να πω πως και η γνωμοδότηση δική μας προσπαθώντας να δώσει μια σύνθεση είναι επίσης ένα περίπλοκο κείμενο να κατανοήσει κανείς. Επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο θα έλεγα τα εξής. Να σας πω πως το βασικό μήνυμα της δικής μας γνώμης για την ίδια την ΚΑΠ ως δημόσιας πολιτικής και το μήνυμα που έχει να κάνει με το μήνυμα που θα φέρει τα παραδοτέα έχει ως εξής. Ο ορισμός για την ΚΑΠ, το πρώτο μήνυμα είναι πως θεωρούμε πως δεν υπάρχει αρκετά σαφές μακροπρόθεσμο όραμα στα πλαίσια αυτής της μεταρρύθμισης. Δεν λέμε πως δεν έγιναν μελέτες, δεν λέμε πως δεν, έγινε, δεν παρουσιάζονται υποθετικά σενάρια. Όχι, πολλά. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι ποια είναι το συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο όραμα το οποίο στηρίζει μέσω των βασικών εναλλακτικών που προσφέρει αυτή η μεταρρύθμιση. Το δεύτερο μήνυμα το εξή. Χρειαζόμαστε ε, στέρεα οικονομικά επιχειρήματα τα οποία δεν έχουν κατατεθεί και κυρίω δεν έχει γίνει για το μεγάλο ρόλο των άμεσων ενισχύσεων. Δεν λέμε πως δεν έχουν συλλεχθεί δεδομένα. Δεν λέμε πως δεν υπάρχουν οικονομικά τεκμήρια. Θεωρούμε όμως πως δεν είναι στέρεα για να ενισχύσουν ε, αυτά τα οποία παρουσιάζονται για το βασικό πυλώνα αυτής της αγροτικής πολιτικής. Το δεύτερο μήνυμα το τρίτο είναι πως οι στόχοι και οι φιλοδοξίες για, τα το περιβάλλον και το κλίμα θα βασίζονται στα κράτη-μέλη, στις προθέσεις τους ε, και στις προτάσεις ε, της Κομισιόν. Και το 30% που θα προσφέρει η ΚΑΠ δεν είναι ρεαλιστικό κατά τη γνώμη μας. Έχουμε κάνει μια αξιολόγηση στα πλαίσια της τρέχουσας ΚΑΠ και των εργαλείων που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα. Τέταρτον, οι κανόνες συγχρηματοδότησης δεν απηχούν την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Και επίσης θεωρούμε πως οι οροφές της πληρωμές για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις θα είναι περιορισμένες εάν αποκλειούν, αποκλείονται από την ΚΑΠ οι πληρωμένες και δωρεάν ε, ε, εργασίες, ε, γεωργικές εργασίες και τα κόστη αυτών. Αυτά. Τώρα, για το μοντέλο που θα παραδώσει τους στόχους της ΚΑΠ και με τα πάρα, πολλά, τις πάρα πολλές αλλαγές που προτείνονται, λέμε τα εξής. Βασίζονται σε τέσσερις έννοιες με τις οποίες συμφωνούμε. Επικορικότητα, απόδοση, απλούστευση, λογοδοσία. Για την επικουρικότητα δεν θα πω τίποτα, ούτε και ε, την απλούστευση, δεν έχουμε χρόνο, αλλά θα πω δύο λόγια για την απόδοση και τη λογοδοσία. Για την απόδοση θεωρούμε πως οι προτάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία για, μια, για ένα σύστημα αποτελεσματικού ελέγχου απόδοσης. Γιατί το λέμε αυτό. Γιατί λείπουν κάποια στοιχεία, κατά τη γνώμη μας. Δεν υπάρχουν σαφείς, συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι στόχοι που να μπορούν να μετρηθούν. Τα μέτρα τα οποία σχετίζονται με τους στόχους επίσης λείπουν και δεν έχουμε λείπει επίσης ένα πλήρες σετ ε, δικτών ε, επιπτώσεων, αποτελεσμάτων και εκρών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρόταση αυτή θα αποδυναμώσει ε, τη λογοδοσία. Και γιατί το λέμε αυτό. Γιατί αναγνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον θα είναι σε θέση να πιστοποιεί την πραγματικότητα ακρίβεια και πληρότητα των λογαριασμών, αλλά δεν θα μπορεί να δηλώσει για το μεγαλύτερο κομμάτι των, ε, των δαπανών εάν οι πληρωμές έγιναν στους δικαιούχους σύνομα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το λέμε αυτό γιατί λέμε πως στον οικονομικό κανονισμό λέει πως οι λογαριασμοί θα συνοδεύονται από τη γνώμη ενός ε, ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα όπου η δαπάνη είναι νόμιμη και ε, κανονική. Και αυτό που βλέπουμε είναι πως έχουμε εδώ δύο διαφορετικούς χώρους δαπάνης. Τις δαπάνες εκτός στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και αυτά τις δαπάνες που βρίσκονται μέσα στο στρατηγικό σχέδιο. Το πρώτο είναι το 2% της δαπάνης για την ΚΑΠ και εκεί κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θα έχουμε την επαλήθευση της νομιμότητας και της κανονικότητας από ανεξάρτητους φορείς. Στο δεύτερο που είναι το 90%, το 98% των δαπανών της ΚΑΠ, αναγνωρίζουμε πως η αξιολόγηση θα γίνεται και αναγνωρίζουμε πως η αξιολόγηση των συστημάτων διαχείρισης θα γίνονται και για τις διαχειριστικές αρχές και για τις βασικές απαιτήσεις. Ναι, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι θα γίνεται επαλήθευση από ανεξάρτητους φορείς για τις πληρωμές που γίνονται στους τελικούς δικαιούχους και αν είναι αυτές σύνομες με την εθνική ε, νομοθεσία. Ε, κάτι το οποίο είναι απέτηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και για το λόγο αυτό λέμε πως υπάρχει μια αποδυνάμωση ε, στο νέο σύστημα στην αρχή της λογοδοσίας. Και σας υπενθυμίζουμε πως έχουμε διεθνή πρότυπα τα οποία λένε πως χρειαζόμαστε διαφόρων ειδών ελέγχους, αλλά επίσης να γίνονται ε, επίσης ε, ε, τεστ ουσιαστικότητας που δεν βρίσκουμε μέσα στο καινούριο σύστημα. Οπότε, Να σας πω γιατί σε εκτός καπ, στρατηγικών σχεδίων πληρωμές δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά για τους τελικούς δικαιούχους δεν θα επαληθεύονται παρά μόνο οι μεταβιβάσεις στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, εμείς χαιρετίζουμε αυτή την μετακίνηση προς μία ε, προσέγγιση που θα μετράει την απόδοση και τη συμμόρφωση, αν είναι στέρεα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ελέγχουμε την νομιμότητα και την κανονικότητα, σύμφωνα με το όσο λένε οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Τσέλε είναι ο εισηγητής μας. Σας παρακαλώ όλους να είστε πολύ σύντομοι. Ναι, σύντομο, Πρόεδρε. Αλλά για το θέμα της αγροτικής πολιτικής υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφέρουμε. Θα προσπαθήσω να τα φιλτράρω κάπως αυτά που θέλω να πω. Υπάρχει, ακούσαμε την ε, θέση του ελεγκτικού συνεδρίου και ευχαριστώ τον κύριο Φιγκερέιντο και του συνεργάτες του. έχουν, ε, μας μίλησαν για προτάσεις για τις μεταρρυθμίσεις της κοινή γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν ε, θετικά στοιχεία σε αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής πολύ συχνά απηχούν ε, και αυτά τα οποία τονίζει το Κοινοβούλιο, ότι θέλουμε μεγαλύτερη απλούστευση των ε, κανονισμών. Θέλουμε ένα σύστημα που να βασίζεται περισσότερο στην απόδοση. Και παράλληλα παρατηρούμε κάτι το οποίο προσπαθήσαμε να επιτύχουμε και στη μεταρρύθμιση στο τωρινό πλαίσιο της στρατηγικής για τη γεωργία. Να έχουμε απλούστευση χωρίς να έχουμε μείωση των ε, ε, ενισχύσεων. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε δηλαδή ε, κάτι άλλο παρά το σύστημα υπολογισμού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να φροντίσει ώστε τα κράτη-μέλη ε, να τηρούν τις διατάξεις. Στο πλαίσιο ε, της εισαγωγής της πράσινης νομοθεσίας του greening είδαμε πολλά εμπόδια και πολλές κριτικές. Ακούσαμε ε, και τα όσα μας είπαν στη διαδικασία της απαλλαγής ότι δεν επετέφθησαν οι στόχοι τους οποίους ε, είχαμε θέσει. Το συνολικό σύστημα υποστήριξης της γεωργίας από πλευράς του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού ε, δεν είναι επικαιροποιημένο. Δηλαδή θέλουμε να υπάρχει καλή απόδοση, καλή παραγωγή και να τηρούνται και κάποια κριτήρια που έχουν σχέση με την αγορά. για το αν οι ενισχύσεις ακολουθούν κάποια έννοια επικουρικότητας ε, και πού απαιτείται κάποια υποστήριξη όταν διαπιστώνουμε ένα είδος βιομηχανοποίησης ε, στη γεωργία ε, το εισόδημα μπορεί να μετρηθεί με ανεπαρκείς μονοτρόπους. Γιατί μπορεί κάποιο να έχει ένα μικρό εισόδημα και από την άλλη πλευρά ε, να έχει μεγάλες άμεσες ενισχύσεις. Σαφώς λοιπόν μπορούμε να διαπιστώσουμε κάτι το οποίο δεν πάει καλά. Ε, για το ερώτημα του τι στόχους θέτουμε για την κοινή γεωργική πολιτική, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους άλλους στόχους για την ευρωπαϊκή πολιτική, για το κλίμα, για το περιβάλλον. Θέλουμε να έχουμε διαφοροποίηση να δούμε σε τι βαθμό αυτό διευκολύνεται από τα κράτη-μέλη κατά πόσο συμβαδίζουν τα κράτη-μέλη δηλαδή και αν μπορεί να επιτευχθεί με κάποια σχέδια στρατηγικής όπου θα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία τίθενται και ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απαντήσει σε κάποια από αυτά τα ερωτήματα. σχετικά με τους στόχους που θέτουμε για την προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και για το αν η νέα στρατηγική μπορεί να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. το capping, ο περιορισμός των ενισχύσεων για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι μια σωστή προσέγγιση, αλλά ήδη από συναδέλφους ακούω ότι είναι αμφιλεγόμενο μέτρο και ελπίζω ότι θα μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η κατάλληλη πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, τουλάχιστον ώστε να σώσουμε αυτά τα οποία πρέπει να διασωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ μια ερώτηση, λέει η Πρόεδρος. Αυτές οι υποκείμενες ε, συναλλαγές που ανέφερε το ελεγκτικό συνέδριο μεταξύ ευρωπαϊκού επίπεδου και επίπεδου κράτους μέλους. Ε, ισχύει αυτό που μας είπαν και τι συνέπειες έχει αυτό και τι γίνεται με το θέμα της ε, regularity και legality των ε, πληρωμών. Έχουμε μια εικόνα του τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος ή ε, δεν έχουμε καθόλου εικόνα. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πολύ σοβαρό. Γι' αυτό θα ήθελα να προσθέσω και εγώ αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Σαβάμα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την γνωμοδότηση αξιότιμα μέλη. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο και την πρωτα... για την πρόταση της Κομισιόν για να σας δώσω τη δυνατότητα να καταλάβετε τα σημαντικά σχόλια που προτίθεμαι να κάνω για την γνωμοδότηση αυτή. Πρώτα απ' όλα Έχω την αίσθηση ότι το πρόβλημα του ελεκτικού συνεδρίου είναι και πάλι η ανάγκη να υπάρχει ένα σωστή, μια σωστή ισορροπία. Μείωση του φόρτου μεταξύ αγροτών και αρχών και το κόστος των ελέγχων και διασφάλιση αποτελεσματικών οικονομικών ελέγχων ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κατάχρηση δημοσίων χρημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε μια έκθεση ιδέα πρωτοβουλία για την προστασία των ιδίων συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων, ε, σε σχέση με περιπτώσεις κατάχρησης στο πλαίσιο τη κοινή αγροτική πολιτική. Ε, ζητήσαμε να υπάρχει μια ΚΑΠ βασισμένη στι στις επιδόσεις και λιγότερο ε, και πιο αποτελεσματική. Πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Φαίνεται ότι ορισμένα από τα σημεία κλειδιά που έθεσε η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού σε εκείνη την έκθεση πράγματι ελήφθησαν υπόψη από την Κομισιόν στην πρόσφατη πρότασή τη, όπω η επέκταση τη χρήση των ενιαίων ελέγχων. Και το λέω αυτό διότι αυτά τα παραλείψατε στην παρουσίασή σα και έχω την αίσθηση ότι θα έπρεπε να υπογραμμίζονται περισσότερο στην γνωμοδότηση. Φαίνεται ότι η προσέγγιση της Κομισιόν όσον αφορά την απλούστευση της ΚΑΠ ήταν να ενδυναμώσει τα κράτη-μέλη, να τα χειραφετήσει και να επικαιροποιήσει το πλαίσιο ελέγχων ώστε να λαμβάνει υπόψη του μεταλλασσόμενου αυτού ρόλου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ το θέμα είναι αλλαγή ρόλων στην όλη πρόταση για την ΚΑΠ και ευθυνών μεταξύ αγροτών, κρατών μελών και επιτροπής. Για να λειτουργεί καλά στο μέλλον η ΚΑΠ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει μια, ένας προσανατολισμός βασισμένος στις επιδόσεις. Οι αρχές να έχουν την ευκαιρία να σχεδιάζουν μέτρα έτσι ώστε να είναι τα καταλληλότερα δυνατά για τι περιοχέ του, για τι περιφερειέ του και για τα κράτη-μέλη. Αν θέλουμε να δούμε αποτελέσματα από αυτό το εγχείρημα, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι η μόνη οδό για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό θα σημαίνει λιγότερο λεπτομερεί ε, νομοθεσίε, αλλά όχι λιγότερου ελέγχου, πιο απλή νομοθεσία, μεγαλύτερη ευελιξία στο σχέδιο, στα εθνικά σχέδια, με μετρήσιμοι στόχοι που να σχετίζονται με τα κονδύλια. Συμφωνώ με το ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει να δούμε κάπως περισσότερο πώς θα ορίζουμε τις επιδόσεις. Αλλιώς θα καταλήξουμε πάλι σε ατέρμονες αναλύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, ατέρμονους ελέγχους που δεν καταλαβαίνει κανείς ούτε ο αγρότης ούτε το κοινό. Στην πρόταση της ε, Κομισιόν φαίνεται ότι η αιτήσια καθάριση επιδόσεων ε, απαιτεί διασφάλιση των υποκειμενών πληρωμών και οι ίδιοι οργανισμοί παρέχουν την ίδια αξιοπιστία, την ίδια διασφάλιση. Θα πρέπει να δίνεται ίδια προσοχή όχι στη συμμόρφωση με λεπτομέρειες, αλλά στα αποτελέσματα. Αντίθετα από την πρόταση της Κομισιόν όμως φαίνεται ότι το ελεγκτικό συνέδριο τώρα καλωσορίζει την εισαγωγή νέων απαιτήσεων που θα πρέπει να ελέγχονται χωρίς να θέλουν να εγκαταλείψουν τις παλιές απαιτήσει. Σίγουρα δεν είχαμε προβλέψει εμεί κάτι τέτοιο στην εκθέση του 2015. Πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι τα πράγματα γίνονται μόνο με έναν τρόπο και ότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο. Ο παλιό τρόπο δηλαδή. Αν ξεκινάμε αυτή την οτροπία, θα καταφέρουμε ποτέ να βελτιώσουμε τι πολιτικέ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη. Είχα μόνο μια πρόταση, λέει ο κύριο Σάβαρο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μάγκελε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Φιγκερέδο, μέλη της Επιτροπής. Τα τελευταία χρόνια επικρίνεται συχνά, δικαίως ή ε, αδίκως, ε, για διάφορους λόγους η ΚΑΠ. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πτυχές, ε, το περιβάλλον και το κλίμα της ΚΑΠ και η κατανομή των τη στήριξη εισοδημάτων, ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της δικαιοσύνης. Και υπάρχει και άλλο ένα θέμα που όλο ένα και πιο επίκαιρο γίνεται, τα παράπονα για την πολυπλοκότητα και το διοικητικό φόρτο λόγω της ΚΑΠ. Πολλές από αυτές τις παρατηρήσεις έχουν γίνει στην ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η Κομισιόν ακούει προσεκτικά οι μεταρρυθμίσει που προτείνονται στην Κομισιόν είναι μια σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπιση ε, των ζητημάτων. Γι' αυτό το λόγο στο περιβάλλον και στο κλίμα έχουμε δώσει περισσότερη έμφαση. Γι' αυτό το λόγο η εισοδηματική υποστήριξη θα πλαισιωθεί καλύτερα με διάφορα μέσα, με ανακατανομή των πληρωμών. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να φύγουμε από το φαύλο κύκλο των όλο και πιο λεπτομερών κανόνων ελέγχων και ελέγχων. Γι' αυτό το λόγο ε, στην πρόταση εστιαζόμαστε στους στόχους και στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Η γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου περιλαμβάνει πολλές επικρίσεις. Για μας αυτό είναι απόλυτα νομιμοποιημένο και αυτό είναι ο ρόλος του ελεκτικού συνεδρίου. Θα διαβάσουμε, θα μελετήσουμε προσεκτικά τη γνωμοδότηση. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Αυτό που μας λείπει είναι ότι κατά την άποψή μας η γνωμοδότηση δεν καταγράφει σωστά την όλη φιλοδοξία της πρότασης ούτε τις πολιτικές και διοικητικές πραγματικότητες. Να σχολιάσω τρία βασικά ζητήματα εισοδηματική υποστήριξη, περιβάλλον και κλίμα και το νέο μοντέλο παράδοση αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τι νέε άμεσε ενισχύσει, η αξιολόγηση επιπτώσεων ε, παρέχει αποτελέσματα για την, υποστήριξη, την εισοδηματική υποστήριξη και την ορίζει ως σημαντικό παράγοντα για τη διατροφική ασφάλεια, τις κλιματικές ε, φιλοδοξίες ε, και τη διατήρηση της υπαίθρου στο μέλλον. Το κάπινγκ, τα ανώτερα επίπεδα, θα βοηθήσουν σε δικαιότερη κατανομή της υποστήριξης. Λέγεται ότι δεν ε, υποστηρίζονται τα περιβαλλοντικά και τα κλιματικά φιλόδοξα σχέδια. Εμείς διαφωνούμε. Ίσα ίσα η πρόταση της Επιτροπής αντιμετωπίζει παλιότερες επικρίσεις του ελεκτικού συνεδρίου, ειδικότερα την έλλειψη της αποτελεσματικότητας του greening, για να αναφέρω μόνο ένα. Η νέα πράσινη αρχιτεκτονική περιλαμβάνει ενισχυμένη ρησιμότητα βάσει Εκταση για όλους τους δικαιούχου ε, χωρίς ε, τις ε, σημερινέ εξαιρεσει. Τα νέα οικολογικά συστήματα, περιβαλλοντικά και κλιματολογικά σχέδια στον πυλώνα 2, δαπάνες στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης με περισσότερους περιορισμούς λόγω της, του αποκλεισμού ενισχύσεων για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, με φυσικά εμπόδια. Το backsliding απαγορεύεται και έχουν συμπεριληφθεί ε, συνδέσεις με την περιβαλλοντική και κλιματική πολιτική. Η πρόταση απαιτεί από τα κράτη-μέλη από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές του αρχές και από την κοινωνία των πολιτών να συμμετέχουν αυτές οι αρχές στην ε, ε, προετοιμασία στρατηγικών σχεδίων για την ΚΑΠ και για άλλα περιβαλλοντικά και κλιματικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ΚΑΠ. Να σας πω και το νέο μοντέλο παράδοσης που κατά την άποψή μας σχετίζεται στενά με τα ουσιώδη κομμάτια της δικών μας προτάσεων πολιτικής. Ε, το Ερεκτικό Συνέδριο έχει καλέσει την Κομισιόν να ενισχύσει τις επιδόσεις της ΚΑΠ. Πολλές από τις ειδικές εκθέσεις τελευταία προτείνουν να δούμε την επίτευξη των στόχων περισσότερο και το πώς επηρεάζει η πολιτική μας τα πράγματα. Αυτό ακριβώ εξετάζουμε εδώ στο νέο μοντέλο παράδοση. Θέλουμε να παρακολουθούμε την επίτευξη στόχων από τα κράτη-μέλη και αυτό να το ενσωματώσουμε στη διαδικασία αξιοπιστία. Να διατηρήσουμε το σημερινά τα σημερινά συστήματα διακυβέρνηση τη ΚΑΠ σε συνδυασμό με πολιετή παρακολουθήσει και καθαρίσει για να αντιμετωπίσουμε τι καταστάσει όπου οι δαπάνε δεν αντιστοιχούν στα αποτελέσματα. Η μηχανική προσέγγιση της γνωμοδότησης όσον αφορά τις επιδόσεις ε, βάσει ευρωπαϊκών στόχων είναι καθαρά τεχνοκρατική και δεν αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική κατά την άποψή μα. Ε, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Όσον αφορά την αξιολόγηση του προτινόμενου μοντέλου αξιοπιστία, ε, μα προβληματίζει η ασάφεια που παρατηρεί το ελεκτικό συνέδριο σε ορισμένου τομείς. Ε, ενώ υπάρχουν σαφείς, σαφείς προτάσεις στην πρόταση. Το νέο μοντέλο αναφέρεται καθαρά στην πρόταση η νομοθεσία τη Ευρώπη θα πρέπει να καθοδηγεί τα κράτη-μέλη για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στου δικαιούχου. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 9 του κανονισμού για το στρατηγικό σχέδιο και στο άρθρα 35 και 53 του οριζόντιου κανονισμού. Το ίδιο ισχύει για το ρόλο των οργανισμών πιστοποίηση, ειδικότερα όσον αφορά τον έλεγχο του κατά πόσο τα συστήματα διακυβέρνηση των κρατών λειτουργούν σωστά. Αυτό περιλαμβάνει έλεγχο τη στήριξη των βασικών απαιτήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κρατη αυτός είναι νόμιμος έλεγχος, ο έλεγχος νομιμότητας και ε, νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών. Τέλος, επιμένοντας την εφαρμογή βασικών κανόνων σε επιμέρους δικαιούχους, η γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου θα οδηγήσει σε ένα διεπίπεδο σύστημα, όπου το υπάρχον επίπεδο συμμόρφωσης με κανόνες επιλεξιμότητας σε επίπεδο δικαιούχων θα συμπληρώνεται από ένα νέο επίπεδο επιδόσεων. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιο επιπλέον φόρτο για όλους τους παράγοντες, πιο αργά παρακαλώ λέει η Πρόεδρος. Ωστόσο το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει σε τεράστιο επιπλέον φόρτο για όλους τους φορείς ε, ήταν ακριβώς ο λόγος που η Κομισιόν προτείνει ένα σύστημα εστιασμένο στις επιδόσεις, κάνοντας μια υποχώρηση σημαντική για τη συμμόρφωση. Η Κομισιόν φυσικά θα λάβει υπόψη τις συστάσεις ε, του ελεγκτικού συνεδρίου για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΚΑΠ και για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους κανόνες. Εδώ εργαζόμαστε βάσει της αρχής ότι τίποτα δεν είναι τέλειο αυτό ισχύει για προτάσεις ε, και για προτάσεις όπως αυτή της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ωστόσο λυπούμεθα που η γνωμοδότηση ε, παραμένει άκαμπτη για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ενώ κάποια ευελιξία θεωρούμε εμείς θα μας βοηθούσε να, για να δημιουργήσουμε μια διαδικασία που θα μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Στις δικές μου ερωτήσεις δεν άκουσα όμως απάντηση. Η πρώτη ερώτηση σχετιζόταν με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Το μοντέλο παραδοσής έχει σχεδιαστεί έτσι που οι ευρωπαϊκοί κανόνες ε, θα αφορούν τα κράτη-μέλη ε, και τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη διακριτική ευχαίρεια που τους παρέχει η πρόταση ώστε να δημιουργήσουν το νομικό πλαίσιο για τους επιμέρους δικαιούχους. Τι θα κάνουμε στο μέλλον. Συνεπώς, και αυτό θα είναι και καθήκον αυτών των οργανισμών πιστοποίηση, θα είναι ότι θα ελέγχουμε κατά πόσο τα συστήματα διακυβέρνηση των κρατών μελών, οι φορεί διακυβέρνηση λειτουργούν σωστά. Μιλάμε για του διαφορού οργανισμού πιστοποίηση, συντονισμού κτλ. Και τέλος, και δεύτερον, τέλος κατά πόσο τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανόνες όταν βρίσκονται ή αν υπάρχουν σωματικέ ελλείψει στα συστήματα διακυβέρνηση και στην εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μου θυμίσετε τη δεύτερη ερώτηση, παρακαλώ. Ποιε είναι αυτέ οι υποκείμενε συναλλαγέ, από ποιον προ ποιον. Το άρθρο 35 του οριζόντιου κανονισμού λέει ότι η επιλεξιμότητα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στο μέλλον θα επηρεάζει τι δαπάνε που δηλώνονται από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι η νομιμότητα και η κανονικότητα, αν ακολουθήσουν οι νομοθέτες αυτή την πρόταση και αποφασίσουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα υπολογίζεται στη σχέση μεταξύ του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους. Δηλαδή, θα ελέγχεται αν κατά την ε, μεταβίβαση 2 δισεκατομμυρίων ε, στο κράτος μέλος έγινε κάποιο σφάλμα ή όχι. Δεν θα ξέρουμε τι γίνεται σε επίπεδο δικαιούχου. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το οποίο περιέγραψα, Πρόεδρε. Δεν έχουμε το χρόνο για να σας τα περιγράψω με κάθε λεπτομέρεια. Α, παρακαλώ, παρακαλώ, έχετε όσο χρόνο θέλετε. Αυτό το οποίο θα ελέγχετε από τα αρμόδια όργανα ελέγχου, που θα είναι ο Οργανισμός Πιστοποίησης και η Επιτροπή, είναι καταρχήν αν τα κράτη-μέλη έχουν ιδρύσει ένα σύστημα ε, ε, ε, σωστής διαχείρισης. Αν υπάρχει μια αρχή διαχείρισης, αν υπάρχουν οργανισμοί πιστοποίησης που λειτουργούν σωστά, αν υπάρχει οργανισμός πληρωμών και γίνεται ορθή εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο θα ισχύσει και για το σύστημα ΟΣΔΕ. Και ένα από τα βασικά ε, σημεία της μεταρρύθμισης, της πρότασης μεταρρύθμισης, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα ε, αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από το πεδίο της δημιουργίας κανόνων. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίζει πολύ λιγότερους κανόνες. Ε, εκεί όπου υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν παράπονα για πολυπλοκότητα και διοικητικό άχθος, δεν θα μιλάμε για το λεπτομερές ε, μήκος και ύψος του φράχτη και της ενδιάμεσης ζώνης. Όλα αυτά δεν θα τα ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε λιγότερες ε, κοινοτικές διατάξεις και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν για τις παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνουν στο πλαίσιο των γενικών γραμμών που θα έχουν θέσει οι κοινοτικοί κανονισμοί και θέτοντας τους κατάλληλους στόχους ούτως ώστε να μπορούν να ελέγξουν ε, οι οργανισμοί πληρωμών αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και θα ελέγξουμε το αν τα κράτη-μέλη ε, συμβαδίζουν με τους, με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν θα γίνεται έλεγχος από την Επιτροπή για κάθε μεμονωμένη υπόθεση για το αν όλο το νομικό πλαίσιο που βασίζεται σε εθνικό δίκαιο ε, συμμορφούνται με, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Διαφορετικά θα είχαμε ένα σύστημα όπου θα είχαμε ε, στοιχεία για την απόδοση με τεράστιες απαιτήσει για την υποβολή εκθέσεων για την απόδοση ε, και άλλο ένα στρώμα που θα αφορά τη συμμόρφωση με όλες τις πολυπλοκότητες του συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα είχαμε υπερβολικά μεγάλο διοικητικό φόρτο και οι νομοθέτες και το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη δεν θα επέλεγαν ποτέ ένα τέτοιο σύστημα. Επιλέγουμε λοιπόν ένα σύστημα που βασίζεται στην απόδοση και πρέπει να γίνει κάποια επιλογή. Σε κάποιο βαθμό κάνουμε πίσω από τον έλεγχο της συμμόρφωσης, κρατώντας βέβαια τις διασφαλίσεις για να ξέρουμε ότι αυτά τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται σε επίπεδο κράτου μέλους ε, όταν εφαρμόζει το κάθε κράτος, μέλο ε, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, για τη θεωρία τα κατάλαβα, λέει η πρόεδρο. Δηλαδή, μεσοπρόθεσμα θα, ε, είναι, θα δούμε το τέλος των γεωργικών ταμείων. Δεν θα υπάρχει κανένα σχετικό σκάνδαλο. Το ελεγκτικό συνέδριο, θέλετε ξανά το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλια. Θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είπε ο κύριος Τσέλερ για την έκθεσή μας σχετικά με το greening και για τις ερωτήσεις που κάναμε σχετικά με το greening. Ε, και άκουσα και τις ερωτήσεις του κυρίου Σάβαμα για τον καλύτερο σχεδιασμό των στόχων. Ευχαριστούμε και την κυρία Γκρέσλε για τις ερωτήσεις της. Είναι πολύ καλές οι ερωτήσεις που έγιναν. Πολύ εύστοχες. Και ακούσαμε και τον κύριο Μαγκάλιο που είπε ότι θα βελτιωθούν ε, τα συστήματα βάσει αυτών των ε, απαιτήσεων. Πιστεύω ότι το θεμελιώδες ερώτημα για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής σας είναι θέματα που αφορούν την ε, λογοδοσία. Θέλουμε μια καλή ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ελέγχου τήρησης του νόμου και θέλω να είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θέλει να υπάρχουν λεπτομερείς κανόνες. Εμάς δεν μας ανησυχούν. Δεν μας ανησυχεί το αν τηρούνται οι λεπτομερείς κανόνες από τους τελικούς δικαιούχους, αλλά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανησυχεί για το αν οι κανόνες που έχουν εγκρίνει οι νομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τηρούνται από τα κράτη-μέλη. Γιατί αν δεν έχουμε έλεγχο αυτών των κανόνων που εγκρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για ποιο λόγο θεσπίζονται αυτοί οι κανόνες. Θέλουμε οι κανόνες να τηρούνται και πρέπει να τους ελέγχουμε για να είμαστε σίγουροι ότι τηρούνται. Οι γενικέ διατάξει, οι γενικοί κανόνε στου οποίου θεσπίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρούνται και αυτό πρέπει να ελέγχουμε. Και το ερώτημα είναι αν σε αυτού του κανονισμού είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Πιστεύω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία για να κρίνουμε ε, ε, το αν τηρούνται όλα αυτά, εάν λειτουργούν καλά τα συστήματα των κρατών μελών. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται σε επίπεδο τελικού δικαιούχου. Δηλαδή, αν οι γενικοί κανόνε στου οποίου εσεί έχετε θεσπίσει το Κοινοβούλιο τηρούνται από του τελικού δικαιούχου. Δεν ζητάμε να πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τον κάθε τελικό δικαιούχο. Ούτε το ελεγκτικό συνέδριο, γιατί αυτό θα ήταν το μεγάλο βάρος των ελέγχων. Αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου σε επίπεδο κράτους μέλους και αυτός ο ανεξάρτητος οργανισμός ελέγχου να μπορεί να δηλώσει ότι οι πληρωμές που γίνονται στους τελικούς δικαιούχους τηρούν τους κανόνες που έχετε θεσπίσει εσείς στο Κοινοβούλιο. Αυτό θέλουμε εμείς. Οι κανόνες που μπαίνουν στα σχέδια σε κάθε κράτος μέλος για τη γεωργική πολιτική θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι δύσκολο να θεσπιστούν τέτοιοι μηχανισμοί που θα έχουν βέβαια κάποιες συνέπειες. Αλλά ούτε ζητάμε επικάλυψη ελέγχων, ούτε μεγαλύτερο διοικητικό άχθος. Αυτό που ζητάμε είναι κάποιος μέσα στο όλο αυτό σύστημα, κάποιος, όχι όλοι μαζί, κάποιος φορέας να κάνει τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας. Ούτω ώστε να ελέγχουμε ότι οι κανόνες που έχει θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το, Ευρωπαϊκό, και το Συμβούλιο τηρούνται. Αν τηρούνται στο επίπεδο κράτους μέλους. η Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους για το αν υπάρχει αυτή η νομιμότητα και η κανονικότητα των διαδικασιών. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ο εισηγητής για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ναι, αυτό το θέμα παραμένει, παραμένει συνεχώς. Το έχουμε συζητήσει. Υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη σε κάθε επίπεδο ότι οι κανόνες που αποφασίστηκαν από όλους μας από κοινού τηρούνται στην πράξη, μεταφέρονται σε εθνικό δίκαιο και τηρούνται. Στο Κοινοβούλιο πολλές φορές ε, θέλουμε να έχουμε κάποια αποτελέσματα από τους πολιτικούς με τους οποίους συζητάμε σε ε, εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα πρέπει να ε, εξασφαλίζει ότι έχει εμπιστοσύνη στους φορείς των κρατών μελών. οι συνάδελφοί μα, στην αρμόδια επιτροπή θα πρέπει επίσης να φροντίσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Καλώ ευχαριστώ. Πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Έχουμε και τους συναδέλφους ε, της Όλαφ ε, και ξέρουμε ότι έχουν πάρα πολλά ευρήματα και πάρα πολλές πληροφορίες ε, φαντάζομαι για διάφορες χώρες, όχι μόνο για μια χώρα. Λίγη η δημόσια συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστούμε για τις διαφωτιστικές παρουσιάσεις σας.